Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας παρακαλώ. Φορέστε τα ακουστικά, εφόσον ε, επιθυμείτε διερμηνία. Και ας ξεκινήσουμε με το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη, την οποία δεν εξαντλήσαμε σήμερα το πρωί. Πρόκειται για τον απολογισμό της αποστολής αντιπροσωπείας ΕΝΒΗ, της Επιτροπής μας δηλαδή, στην Πολωνία. Πήγαμε λοιπόν στην Πολωνία. Λάινερ, Μακολάτη, Μακίβαν και Χίμπνερ. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω λιγάκι τι έγινε εκεί και θα ακούσουμε μετά και τους συναδέρφους. Η Πολωνία αναλαμβάνει την Προεδρία μετά την Ουγγαρία για την εξάμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό την 1η Ιουλίου του 2011. Κατά το διάστημα αυτό θα υπάρξουν διάφορες εκδηλώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή κατά τη διάρκεια δηλαδή της Πολωνικής Προεδρίας. Η Επιτροπή μας έστειλε λοιπόν μια αντιπροσωπεία στην Πολωνία. Συναντήσαμε εκπροσώπους της πολωνικής κυβέρνησης, ε, εκπροσώπους ε, των δύο σωμάτων της Βουλής, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και δημοσιογράφους. Μιλήσαμε για προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας, όσον αφορά δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 2011. Ειλικρινά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους αφετριονές μας. Μας υποδέχτηκαν πολύ θερμά, μας έδωσαν διάφορες πληροφορίες. Η φιλοξενία τους ήταν υπέροχη. Οι συζητήσεις μας ήταν ιδιαίτερα καρποφόρες. Συζητήθηκαν, συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Η Πολωνία λοιπόν ετοιμάζεται για την Προεδρία της και στον τομέα του περιβάλλοντος, ε, δημόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών. Η αντιπροσωπεία μας διαπίστωσε ότι η Πολωνία εταίροι μας συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και είναι αποφασισμένοι να πετύχει η εξάμεινη προεδρία τους. Ποια ήταν τα κύρια σημεία λοιπόν, τα σημεία κλειδί όσον αφορά την Πολωνική Προεδρία, θέματα δηλαδή που εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Ήταν τα βιοκτώνα, ε, τα απόβλητα και απορρίμματα από ηλεκτρικά είδη, όπως επίσης πηγές ενέργειας και πρόγραμμα εργασιών, ο χάρτης. Όπως αυτός υιοθετήθηκε πρόσφατα. για μια οικονομία δηλαδή όπου η κατανάλωση διοξιδίου του άνθρακα και εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα μειωθούν. Γίνονται προετοιμασίες για τη διάσκεψη κορυφής στο Ρίο Ντετζανέιρο επίσης και συζητήσαμε και γι' αυτό. Τώρα ένα θέμα το οποίο θα είναι ανοιχτό κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας είναι το θέμα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και η μεταρρύθμιση της κοινή ζωικής πολιτικής. Τα μέλη της αντιπροσωπείας διαπίστωσαν ότι οι Πολωνοί εταίροι μας θέλουν να συνεργαστούν στενά με την δικιά μας την Επιτροπή. Μας το είπε αυτό δηλαδή η Πολωνική Προεδρία. Έτσι λοιπόν, Αυτά είχα να πω εγώ αρχικά για την επίσκεψη αυτή. Τώρα ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαρίστω να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια. Χίπνερ και Μάρκουν Λάιτερ μετά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους συναδέρφους που αφοσίασαν το χρόνο τους και αφιέρωσαν το χρόνο τους κατά τη διάρκεια εκείνης της τυρκουάς εβδομάδας με την επίσκεψή μας στην Πολωνία. Γιατί πηγαίνοντας στην Πολωνία δεν μπορούσαν να βρίσκονται στις εκλογικές τους περιφέρειες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά. Όπως είπε και ο πρόεδρος μόλις τώρα, συναντηθήκαμε με τρεις υπουργούς πρώτα απ' όλα. Υγείας, και η υπουργό μας ανέφερε τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Ένα από τα θέματα είναι η γύραση του πληθυσμού. Μας ανέφερε επίσης τα θέματα που σκοπεύει να προτείνει. Επέστησε την προσοχή μας, κατά τα άλλα, και στην ειδική κατάσταση που αφορά τα μικρά παιδιά, τα νήπια. Και μας είπε ότι και αυτό είναι προτεραιότητα για την Πολωνική Προεδρία. Είναι ένα θέμα που είναι και δικιά μας αρμοδιότητας, μια που συζητάμε για διάφορα προϊόντα που κυκλοφορούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απευθύνονται στα μικρά αυτά παιδιά. Πρέπει να φροντίσουμε για την προστασία των παιδιών, όπως επίσης και για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Ο δεύτερος υπουργό με τον οποίο βρεθήκαμε ήταν ε, του περιβάλλοντος. Συζητήσαμε μαζί τα θέματα που μας απασχολούν ε, και μας η ανακύκλωση και η διάρκεια ζωής των προϊόντων. Προτάθηκε ότι ίσως θα έπρεπε να προσφέρουμε νομικές λύσεις για να παρατείνεται η ζωή του οικιακού εξοπλισμού. Γιατί τι γίνεται σήμερα, χρησιμοποιούμε και αλλάζουμε πολύ γρήγορα μηχανήματα. Είναι θέμα λοιπόν ε, ε, καταρχήν εξοπλισμού και δεύτερον ανανεώσιμης ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως θα έπρεπε να προτείνει κάτι στο Ντέρμπαν. Συναντηθήκαμε επίσης και με τον Υπουργό Γεωργίας. Ο Υπουργός Γεωργίας μας μίλησε Κυρίω για την μεταρρύθμιση τη κοινή γεωρικής πολιτική και για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Ανέφερε κάποιε απειλέ που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση. Διότι αν κάθε χώρα μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρει τι δικέ της αποφάσει για ε, του γενετικά τροποποιημένους οργανισμού και του εφαρμόσει στη δικιά τη επικράτεια, αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί αυτοί τελικά θα μετακινηθούν πολύ εύκολα από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι λοιπόν, ε, γιατί το ξέρουμε ότι είναι εύκολο μέσω διαδικτύου να γίνουν τέτοιες προμήθειες. Έχουμε μια ελεύθερη αγορά, άρα πώς θα ελέγξουμε πλήρω το τι γίνεται με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και κατά πόσο αυτοί μεταφέρονται από τη μία χώρα στην άλλη. Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση ήταν επίσης και αυτή που είχαμε με την Επιτροπή Γεωργίας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Οι Πολωνοί συνάδελφοι εξέφρασαν τις δικές τους ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα εκπροσωπήσει στο Δέρμπαν η Πολωνία τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο μας είπανε και για τις τιμές της ενέργειας και κυρίως του ηλεκτρισμού. Ανέφεραν και τις ανησυχίες τους για το εμπόριο, ε, για το εμπόριο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σύνορα θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί και αυτό το θέμα. Συναντηθήκαμε και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όπω συμβαίνει συνήθω σε τέτοιε συναντήσεις, έτσι και αυτή τη φορά, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον μίλησαν κυρίως για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μας ανέφεραν θέματα λοιπόν προστασίας του περιβάλλοντο μέσα στα οικονομικά πλαίσια που βρισκόμαστε. Συναντηθήκαμε και με τα μέσα ενημέρωση με δημοσιογράφους, ε, συνέντευξη τύπου που δώσαμε. Οι ερωτήσει του όμω ήταν ε, λίγες, οι ειδικέ ερωτήσεις. Ο πρόεδρο μα προσπάθησε να τους παρουσιάσει τα επιτεύγματά μας. Προσπάθησε να τους παρουσιάσει με ποιο τρόπο καταλήγουμε σε συμπεράσματα από κοινού, σε συνεργασία βέβαια με το Συμβούλιο. Ήταν πάντω σαφέ ότι δημοσιογράφοι και όχι μόνο η Πολωνοί αλλά και άλλοι που είναι διαπιστευμένοι στην Πολωνία δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά πώς είναι η δομή, η διάρθρωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων τώρα που έχουμε περάσει στις διαδικασίες της συνθήκης της Λισαβόνας. Είμαι σίγουρη ότι και άλλοι θα το πούν ότι μιλήσαμε και για την πυρηνική ενέργεια. Δεν θα πω εγώ σε λεπτομέρειες γι' αυτό. Απλώς θα σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να σας πω ότι πιστεύω πως η συνάντηση αυτή στην Πολωνία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ελπίζω να σας άρεσε η Πολωνία. Ελπίζω να περάσατε καλά και την επόμενη φορά που θα πάμε στην Πολωνία να είμαστε ακόμα περισσότεροι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Φίτνερ. Ραλβίλα Μαρτνέιτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την προετοιμασία, την επιτυχή προετοιμασία αυτή τη επίσκεψη και επίση ευχαριστούμε και του συναδέλφου για την υποδοχή που μα επιφύλαξαν. Πριν από την ε, ανάληψη τη Προεδρία, είναι πάντοτε χρήσιμε τέτοιε επισκέψει σε τέτοιε χρονικέ συγκυρίε. Βεβαίω, είναι καλό να μαθαίνει επίση κανεί ποιε είναι οι προτεραιότητε τη κάθε Προεδρία. Συναντήσαμε, όπως είπατε, τον Υπουργό Υγείας, συζητήσαμε για την ποιοτική παιδική ηλικία, αλλά βεβαίως πρέπει να μας απασχολήσει η υγεία καθόλου των δύο των ε, πολιτών, του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Συζητήθηκαν θέματα σε σχέση με τις ειδικέ ανάγκες που μπορεί να αφορούν ιδιαίτερα στα παιδιά. Ε, όλα αυτά μας απασχόλησαν ιδιαίτερως. Επίσης μιλήσαμε για προγράμματα πρόληψης και για το πώς μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους τα κράτη-μέλη. Στη συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος εκφράσαμε τη θέση μας σε σχέση με τη ρήπανση της Βαλτικής θάλασσας. Από άποψη και περιφερειακή και ευρωπαϊκή, το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όπως είπε και η συνάδελφο. μας απασχόλησε και η πυρηνική ασφάλεια. Θα πρέπει για όλα αυτά τα ζητήματα να μπορούμε να μιλήσουμε με φωνή ενιαία, έχοντας υπόψη ότι ναι, οι πυρηνικοί σταθμοί χτίζονται στα σύνορά μας. Ευχαριστώ πολύ για τη μαρτυρία σας. Περνάμε στο επόμενο λοιπόν σημείο. Ακρόαση για τη Βαλτική θάλασσα. Σας ανακοινώνω ότι αύριο στις 9.30 υπάρχει από τις 9.30 στις 11.30 ούτως ή άλλως ακρόαση για την διαρροή άνθρακα στην κεντρική Ευρώπη. Το Ευρωκοινοβούλιο θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε αυριανή κρόαση. Τώρα, σήμερα θα μας απασχολήσει το θέμα της Βαλτικής και σε σχέση με την βιώσιμη γεωργία. Οι προσκεκλημένοι μας βρίσκονται στην αίθουσα. Να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή. Την εισαγωγή θα κάνουν οι κυρίες Σάτου Χάση και Άννα Ρόσμπαχ και ο κύριος Ολένιτσακ. Η κυρία Σάτου Χάση. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επιτροπή Περιβάλλοντος που διοργάνωσε την παρούσα ακρόαση. Η Βαλτική θάλασσα είναι από τα πιο ε, σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα της χώρας μου που βεβαίως βρέχεται από τη Βαλτική. Συχνά όταν οι Φιλανδοί μιλούν για την θάλασσα εννοούν, όταν λένε θάλασσα δηλαδή εννοούν τη Βαλτική διότι όλη βέβαια η ακτογραμμή μας είναι η ακτογραμμή της ε, Βαλτικής. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Βαλτική δεν αποτελέσε και τόσο πολύ θέμα. Εγώ παρατήρησα ότι υπάρχουν πολλές και πολλοί συνάδελφοι που δεν γνωρίζουν ορισμένα βασικά πράγματα τα οποία ωστόσο είναι κοινή γνώση στην χώρα μου. Η Βαρτική μετά την διεύρυνση της ε, περασμένης δεκαετίας έχει γίνει πλέον στην ουσία εσωτερική ευρωπαϊκή θάλασσα ένα μικρό μέρος της ακτογραμμής ανήκει στην Ρωσία αλλά οι υπόλοιπες χώρες που την περικλείουν είναι, ευρωπαϊκές, είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ό,τι θίγει τη Βαλτική θίγει την Ευρώπη. Η... Άνθρωποι και δικαίως θεωρούν ότι η προστασία του περιβάλλοντος στη Βόρεια Ευρώπη είναι σχετικά σε υψηλό επίπεδο, ε, οι άνθρωποι είναι νομοταγείς και το καθεξής. Ίσως λοιπόν αποτελέσει έκπληξη για σας να σας πω ότι η Βαλτική στο βορρά της Ευρώπης είναι από τις πιο μολυσμένες περιοχές του κόσμου. Ένας από τους λόγους που το εξηγεί αυτό είναι το γεγονός ότι η θάλασσα είναι σχετικά ρηχή με μέσο βάθος μόνο 57 μέτρα. Ενώ για παράδειγμα η Μεσόγειος έχει ένα μέσο βάθος του στάξου του ενός χιλιόμετρου. Είναι λοιπόν μεγάλη, εκτεταμένη θάλασσα, αλλά αλλά δεν μπορεί κανείς να κρίνει τον όγκο των ε, υδάτων της θάλασσας αυτής ε, μόνο εξετάζοντα το χάρτη, γιατί είναι ρηχή θάλασσα όπως είπα. Μιλώντας για μόλυνση, οι περισσότεροι, στο, το μυαλό των περισσότερων ανθρώπων πηγαίνει σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και αυτό είναι δικαιολογημένο εν μέρη όπως έδειξαν οι συζητήσεις που έγιναν σήμερα το πρωί για την περιεκτικότητα των ψαριών της Βαλτικής σε διοξίνες και ιδίως τον Σολομό. Χρειαζόμαστε λοιπόν λήψη μέτρων για να μειωθούν οι επικίνδυνες ουσίες και το πετρέλαιο αλλά το μεγαλύτερο ε, πρόβλημα για την Βαλτική είναι η ευτροφία στον βυθό. Ένα τέτοιο σημάδι είναι ότι είναι μια, μεγάλες περιοχές οι οποίες στερούνται οξυγόνου στα νερά. Στη Βαλτική σημειώνεται αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη θάλασσα του κόσμου. Η ευτροφία στην επιφάνεια σημαίνει για παράδειγμα τοξικά πράσινα, κιανοπράσινα μάλλον φύκια. Μια άλλη έκπληξη για πολλές και πολλούς συναδέλφους είναι ότι ο μεγαλύτερος λόγος που προκαλεί την ευτροφία αυτή είναι εκκλήσεις αζότου και φωσφόρων από γεωργικές καλλιέργειες σε χώρες μέλη της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται σημαντική αλλαγή στις πολιτικές αυτές, στις ε, αγροτική πολιτική δηλαδή, εάν θέλουμε να σώσουμε την Βαλτική. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να σταματήσει η γεωργική εκμετάλλευση, αλλά πρέπει να γίνει με ευφιέστερο τρόπο. Είναι ενδιαφέρον και σημαντικό ότι την επόμενη Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών αναλαμβάνει η Πολωνία με, στα πλαίσια της, στρατηγικής, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ε, Βαλτική έχει συμφωνηθεί η Φιλανδία και η Πολωνία να αναλάβουν τα ενία της ε, αυτή ε, πορείας αυτής. Η νέα φιλανδική κυβέρνηση η οποία πρόκειται να οριστεί τούτη την εβδομάδα και εγώ μάλιστα ήμουν και μία από τις διαπραγματεύτριες του κυβερνητικού προγράμματος έχει ως ξεκάθαρη εντολή να μειώσει την ευτροφία της Βαλτικής από τα απόβλητα της ε, γεωργίας. Και αυτό θα είναι ένα από τα κέρια θέματα της ε, φιλανδικής θέσεως για την κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την ε, διοργάνωση της παρούσας ακροάσεως και ευχαριστώ και όλες και όλους τους προσκεκλημένους. Ελπίζω ότι τα όσα θα ακούσουμε θα βελτιώσουν και θα αυξήσουν τις γνώσεις μας για το θέμα, ότι θα βοηθήσουν να αναπτυχθεί η σκέψη μας, να εξελιχθεί η σκέψη μας, να προκαλυφθεί και μια ε, αλλαγή νοοτροπίας με ε, απότερο στόχο να γίνει καθαρότερη και υγιέστερη η Βαλτική θάλασσα. Ευχαριστώ κύριε Χάση. Η κυρία Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα δανέζικα. Να ευχαριστήσω πρώτα την κυρία Χάση για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία που ανέλαβε και που νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία. Εγώ προέρχομαι από άλλη χώρα που βρέχεται από τη Βαλτική, από τη Δανία. Όπως είπε η κυρία Χάση, το σύνολο της Βαλτικής ε, είναι μια θάλασσα που υπάρχει από την προϊστορία το νερό κυκλοφορεί είναι πολύ εύκολο να μολυνθεί η θάλασσα αυτή με τα κιανοπράσινα φύκια και να πάσχει τώρα από Στην οικογένειά μου όλοι ήταν ψαράδες. Εγώ στην ουσία γεννήθηκα κάτω από το ψαράδικο ε, σκάφος μας και έχω παρακολουθήσει όλη την εξέλιξη από τα πιο μικρά μου χρόνια. Εκεί έρχονται, ε, ε, στις περιοχές μας έρχονται τα ψάρια για να οτοκίσουν τα μικρά ψαράκια μετά αναπτύσσονται στα πιο θερμά νερά και μεγάλος αριθμός ψαράδων πηγαίνουν στις περιοχές αυτές με μικρούς στολίσκους αλλιευτικών σκαφών αλλά όλες αυτές οι περιοχές έχουν υποστεί τα αποτελέσματα, τα αρνητικά αποτελέσματα των ε, χημικών βιομηχανιών αλλά και ε, των πυρηνικών σταθμών που ψύχονται με θαλασσινό νερό ανεβάζοντας έτσι την θερμοκρασία του περιβάλλοντος θαλάσσιου ύδατος κατά τουλάχιστον 10 βαθμούς. Τέλος πάντων τα μικρά ψάρια τα, τα τρώνε τα μεγάλα, τα μεγάλα συγκεντρώνουν στο ε, λίπος τους τα διάφορα τοξικά στοιχεία και καταλήγουν εν τέλει στο πιάτο μας. Σε ό,τι με αφορά, πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Ακόμα και αν ακόμα και για κάποιον που δεν ενδιαφέρεται πάρα πολύ για θέματα περιβάλλοντος, γιατί είναι εν τέλει θέμα υγείας. Και τουλάχιστον αυτή τη στιγμή αντιληφθούμε ότι είναι θέμα υγεία, θα πρέπει να προξενήσει έντονο το ενδιαφέρον μας. Ορισμένε από τις χώρε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε και η κυρία Χάση, όλες οι χώρες που βρέχονται από την Βαλτική είναι στην ουσία μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεργαστούν για μια πραγματική στρατηγική για την διάσωση της Βαλτικής. Εγώ νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και κινούμαστε ήδη τα τελευταία 10 με 12 χρόνια προς την σωστή κατεύθυνση. Έχουμε σημειώσει πρόοδους, έχουν ληφθεί μέτρα, έχουν επιβληθεί μέτρα τα τελευταία 30 χρόνια, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις των ε, φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων κλπ. στη θάλασσα και επομένως στην υγεία μας. Αλλά δεν έχουμε κάνει όλα όσα θα έπρεπε. Το είπε και η κυρία Χάση αυτό. Πρέπει να τροποποιηθεί και η χρήση ορισμένων ε, γεών γύρω από τη θάλασσα. Πρέπει να θεσπίσουμε ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας. Από το 2003 έχουμε ένα 7% ε, των γεών αυτών που έχουν τεθεί σε καθεστώς αγρανάπαυσης. Χρειάζεται να προστατεύσουμε επίσης ε, τα ποτάμια, δηλαδή τα γλυκά νερά που καταλήγουν στη θάλασσα, ε, τον υδάτινο ορίζοντα και ούτω Τα, τα μέτρα αυτά βέβαια δεν είναι επαρκή ακόμη. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί υπάρχει και το Nord Stream, ο αγωγός Nord Stream δηλαδή που ε, θα ε, κατασκευαστεί αλλά υπάρχει και ένας αριθμός ε, εκρηκτικών βομβών και ούτω καθεξής που έχουν καταλήξει στα βάθη της θάλασσας αυτής και δεν έχουν ακόμα εκραγεί ή δεν έχουν ευτυχώς μέχρι τώρα εκραγεί. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος, κανείς εδώ που να μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Ελπίζω πάντως ότι θα διεξαχθεί εδώ μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Ροσμπαχ. Ο τρίτος άνθρωπος είναι ο κύριος Ολέσνιτσακ πρώην Υπουργό Γεωργία τη Πολωνία. Έχετε το λόγο, αγαπητή κυρία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και ευχαριστώ και για την εξαίρετη αυτή πρωτοβουλία. Ήμουνα εισηγητής για την ε, εφαρμογή της στρατηγικής για την περιφέρεια της Βαλτικής. Γι' αυτό λοιπόν και έχω μερικά σχόλια να σας κάνω. Δουλεύοντας ε, πάνω στην έκθεση αυτή με τους συναδέρφους μου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα μετά από τις παρατηρήσεις μας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την κατάσταση που επικρατεί στην Βαλτική περιοχή. Η Βαλτική περιοχή είναι πολύ σημαντική και για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στα πλαίσια της συνύπαρξης και από κοινού δράσης όλων αυτών που ζουν γύρω από τη Βαλτική θάλασσα. Η Βαλτική λοιπόν στην πραγματικότητα είναι περίπου εσωτερική θάλασσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποτελεί ένα στοιχείο ενωτικό που ενώνει δηλαδή τις χώρες που βρίσκονται γύρω από αυτήν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει. Δεν είναι μεγάλη η Βαλτική θάλασσα, είναι ρηχή και αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τα επίπεδα ζωής στις χώρες που βρίσκονται γύρω από τη Βαλτική θάλασσα. Η στρατηγική λοιπόν για την Βαλτική εκπονήθηκε ακριβώς για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πρώτα απ' όλα έχουμε την προστασία του περιβάλλοντος και έπειτα έχουμε και τις εξελίξεις όσον αφορά την εφημερία. Έπειτα θέλουμε μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης στην περιοχή αυτή και αυτό είναι κάτι που κοιτάξαμε να λύσουμε. Βλέπετε είναι πολύ ελκυστική η περιοχή αυτή, τραβάει τουρισμό. Επίσης έχει και πολλές δραστηριότητες, επιστημονικές, πολιτιστικές. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε τρόπους για συνεργασία μεταξύ των χωρών στην περιοχή. Πρόκειται για 100 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν γύρω από τη θάλασσα αυτή. Οι απειλέ είναι πολλέ. Γι' αυτό ένα άλλο στοιχείο στην έκθεσή μας ήταν και το θέμα της ασφάλειας. Αναφερθήκατε πριν στις χημικές ουσίες. Έχουμε το Nord Stream, τον αγωγό, όπως είπαμε, που επίσης μπορεί να αποτελέσει κάποια απειλή. Γι' αυτό και η στρατηγική μας εκπονήθηκε με, υπό το πρίσμα μάλλον της προστασίας της περιοχής από διάφορες απειλές. Πώς δηλαδή σε περίπτωση κρίσης θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση ή πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε προληπτικά μέτρα για να μην φτάσουμε ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση. Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι η στρατηγική μας αποτελεί ένα πολιτικό άγγραφο. Παρ' όλα αυτά, στην πράξη δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή δεν έχουμε προπολογισμό καταρχήν δεν έχουμε επιμέρους δραστηριότητες και καθήκοντα ε, τα οποία να χειριζόμαστε εμείς από τις Βρυξέλλες. Και αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική αποτελεί ένα σύνολο μέτρων τα οποία μένει να εφαρμοστούν από τα επιμέρους κράτη-μέλη. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, δεν φτάνει. Είχαμε όμως συζητήσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς όμως να ληφθεί τελικά καμία απόφαση που να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την περιοχή αυτή από εδώ. Είπαμε ότι πρόκειται για την εφαρμογή επιμέρους προγραμμάτων από τις διάφορες χώρες μέλη εκεί. Εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε μόνο μέσω της πολιτικής συνοχής. Τώρα υπάρχει συνεργασία μεταξύ τομέων. Η Γεωργία, για παράδειγμα, όμως δεν έχει πετύχει τους στόχους που έχουμε βάλει. Άρα λοιπόν πρέπει να εφαρμοστούν διάφορα μέτρα στο μέλλον, ώστε η στρατηγική αυτή για τη Βαλτική να τεθεί σε εφαρμογή όχι μόνο στον τομέα της συνοχής αλλά και στον τομέα της γεωργίας, της αλίας, του τουρισμού και των υποδομών. Επί του παρόντος δεν βλέπουμε να υπάρχει τέτοιος ε, συντονισμός στο επίπεδο που θα έπρεπε. Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και σε κάτι ακόμα. Θέλω να σας πω ότι ευχαρίστως άκουσα τις απόψεις σας. Είμαι όμως μέλος και της Επιτροπής Γεωργίας και γνωρίζω ότι πολλές φορές υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις προσδοκίες του κόσμου και των κυβερνήσεων. Ίσως και η πολωνική κυβέρνηση να έχει τις δικές της απόψεις. Πολλές φορές ακούμε πόσο πολύ χρειάζονται ε, τα λοιπάσματα, αλλά ακούμε ότι πρέπει να περιοριστεί η χρήση τους. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε και για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, ε, πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά τα θέματα, πάντα όμως με γνώμονα το μέλλον και τις αποφάσεις που θα πρέπει να λυθούν για το μέλλον. Σήμερα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα πάρουν τις ενισχύσεις τους οι αγρότες, πώς θα τους βοηθήσουμε. Να τους βοηθάμε πάντα ε, έχοντας κατά νου την προστασία του περιβάλλοντος. Αν αποφασίσουμε ότι θα πληρώσουμε τα ποσά που έχουν υπολογιστεί βάσει της έκτασης που χρησιμοποιεί ο κάθε γεωργός, αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο, απευθείας. Αλλά οι αγρότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την έκταση, πρέπει να έχουν υπόψη τους και άλλους στόχους που είναι υπέρ του κοινού συμφέροντος. Για την περιοχή λοιπόν της Βαλτικής και τις υποδομές πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν μιλάμε μόνο για επενδύσεις και προγράμματα κοινών επενδύσεων εξαιτίας της γεωγραφικής εγκύτητας, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και πιο μακροπρόθεσμα τις προοπτικές μας. Να δούμε που υπάρχουν και που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, επεξεργασίες αποβλήτων, για παράδειγμα. Να ξέρουμε ότι αν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση πρέπει να καλύπτει όχι μόνο μία πόλη αλλά και άλλες πόλεις, στην Πολωνία για παράδειγμα. Διότι υπάρχουν και άλλες περιοχές που έχουν ποτάμια τα οποία εκκίνονται στη Βαλτική. Άρα και αυτές πρέπει να λυθούν υπόψη και η δικιά τους η πολιτική. Η στρατηγική πάντως και δικιά μου η έκθεση επικεντρώνεται στο θέμα της συνεργασίας με τους γειτονές μας, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία. Χρειάζεται αυτή η συνεργασία. Πρέπει να βρούμε κοινά πλαίσια συνεργασίας. Αλλιώς οι προσπάθειές μας θα είναι ανεπαρκείς. Συχνά τα κονδύλια που δίνουμε για τη συνεργασία χάνονται αν δεν υπάρξουν αντίστοιχε δράσεις και από την άλλη μεριά των συνόρων. Αν δεν υπάρχουν επενδύσεις δηλαδή και εκεί αντίστοιχε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε και να περάσουμε στο πρώτο σημείο της ακροασής μας, που είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Βαλτική Θάλασσα. Εδώ δεν έχω αλλάξει ιδιαίτερα το πρόγραμμα, κάτι μικρό μόνο. Η κυρία Ιωάννα Health θα πάρει το λόγο πρώτα, που είναι υπεύθυνη για την ε, περιφερειακή πολιτική και την ε, πολιτική συνοχής από την μόνιμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το λόγο. Για 7 λεπτά παρακαλώ μόνο. 7 λεπτά παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για την αλλαγή στο πρόγραμμα, αλλά πραγματικά σε 10 λεπτά το πολύ πρέπει να φύγω. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι συνοπτική. Θα σας παρουσιάσω τα σχέδια της ε, Πολωνικής Προεδρίας για την αναθεώρηση της πολιτικής για την πολιτική θάλασσα. Ενώ η συνάδελφος θα μιλήσει για περιβαλλοντικές πτυχές που αφορούν αποκριστικό στη στρατηγική. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον ε, πρόεδρο που μας έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα σχέδια της Πολωνικής Προεδρίας, διότι όπως θα γνωρίζετε, η Πολωνία έχει ιδιαίτερη ευθύνη εφόσον η αναθεώρηση της στρατηγικής ε, επισυμβαίνει στη διάρκεια της Προεδρίας μας, το δεύτερο εξάμεινο της φετινής χρονιάς. Διανύουμε μια ιδιαίτερη χρονική περίοδο, διότι έχουν περάσει δύο, δύο περίπου χρόνια από την πρώτη φάση υλοποίησης της στρατηγικής αυτής θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα δύο τελευταία χρόνια ήταν ένα καλό τεστ, μια καλή δοκιμασία για τον συνολικό μηχανισμό της στρατηγικής και για τους ε, μπλεκομένους, τους εταίρους μας εδώ, που πρέπει να καθορίσουν τους ρόλους τους, τις πρώτες τους δράσεις, δραστηριότητες και να αρχίσουν να υλοποιούν τα ανάλογα προγράμματα. Γι' αυτό νομίζω τη χρονική στιγμή αυτή είναι ε, η καταλληλότερη για να δούμε και να περάσουμε σε αυτή την αναθεώρηση. Λίγα λόγια για το τι ακριβώς είναι η αρμοδιότητά μας εδώ. Υπάρχουν συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίνουν, θεσπίζουν μάλλον τη στρατηγική αυτή από τον Οκτώβριο του 2009 κατά τη Σουηδική Προεδρία. Τότε όντως εγκρίθηκε η στρατηγική αυτή και με το κείμενο αυτό τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο ως το τέλος Ιουνίου 2011 την πρώτη έκθεση πρόοδου. Η έκθεση αυτή πρόκειται να δημοσιευτεί ακριβώς αυτή την εβδομάδα, τις επόμενες μια-δυο μέρες. Ωστόσο, ήδη είχαμε μια προκαταρκτική έκθεση από το Δεκέμβριο του 2010 όπου αναφέρεται ότι οι πολιτικές συζητήσεις θα πρέπει να επιταχυνθούν κατά την Πολωνική Προεδρία και να αποτελέσουν βάση για την αναθεώρηση της στρατηγικής. Γι' αυτό ακριβώς η Πολωνική Προεδρία θα ετοιμάσει το κατάλληλο πλαίσιο για να διεξανθούν οι πολιτικές συζητήσεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ανασυστήσει την ομάδα φίλων της Προεδρίας που είχε δημιουργήσει η Σουηδία όταν είχε αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τις συζητήσεις αυτές θα επικεντρωθούμε στη στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα αυτή καθεαυτή και δεν θα δούμε την ευρύτερη έννοια των στατικικών για μακροπεριφέρειες, μεγαλύτερες δηλαδή γεωγραφικές ζώνες. Εδώ θα χρειαστούμε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως το τέλος τουλάχιστον του 2013 για, την, τον υπολογισμό της προστιθέμενης αξίας των μακροπεριφερειών και ανάλογα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρινούν τη στρατηγική του Δούναβη. Εμεί λοιπόν θα επικεντρωθούμε μόνο στη στρατηγική για την Βαλτική και ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποια προπαρασκευαστικά βήματα, ήδη από την αρχή τη χρονιά. Διοργανώσαμε τον Μάιο διαβουλεύσεις και σε εθνικό επίπεδο αλλά και με συμμετοχή άλλων κρατών μελών Και εδώ είχαμε κάτι μέλη όχι μόνο από τις ε, περιφέρειες των χωρών που βρέχονται από τη Βαλτική, αλλά και εκτός. Ε, σε πρώτη φάση θέλαμε να υποβάλουμε κάποιες νέες ιδέες. Ιδέες της Πολωνίας για την αναθεώρηση, για να δούμε τα θεματικά ζητήματα τι θεματικέ ενότητε που θα μπορούσαν να αποτελέσουν είτε αντικείμενο είτε βάση για την ε, στρατηγική. Επίση, θέλαμε να βολιδοσκοπήσουμε τι προσδοκίε των κρατών μελών σε σχέση με τα θέματα αυτά. Όπω βλέπετε, συνεργαζόμαστε ενεργά και με το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι η πρώτη μα συμμετοχή σε ακρόαση. Την πρώτη ακρόαση για την Ευρώπη τη Βαλτική ε, την πραγματοποιήσαμε στην ε, αρμόδια ομάδα πριν από ένα μήνα το ανάλογο Intergroup και πολύ συχνά πηγαίνουμε και στην Επιτροπή των Περιφερειών για να ακούμε και την άποψη των ε, τοπικών αρχών και των υπευθύνων τους. Πάντως, όπως είπα, η βάση μας ήταν η πρώτη έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποτελεί μάλλον τη βάση μας η έκθεση αυτή μόλις δημοσιευτεί και από τη μέτρηση της πρόοδου θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα από τα δύο χρόνια υλοποίηση της στρατηγική. Πιστεύω ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή θα μας δείξει τι πάει καλά με την όλη στρατηγική και τι επιδέχεται βελτίωση. Πάντως, Εάν δούμε τι συζητήθηκε στι διαφουλεύσει, κάποια από τα σημαντικότερα ζητήματα, κάποιε θεματικέ ενότητε προκύπτουν ήδη από αυτέ τι ε, πρώτε συζητήσει. Η γενική εντύπωση είναι ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διακυβέρνηση και το σύστημα υλοποίησης της στρατηγικής παρά στο περιεχόμενο το ίδιο του προγράμματος δράσης. Τα ζητήματα κλειδιά που έχουν ήδη επισημάνει οι συνομιλητές μας κατά τις διαβουλεύσεις ήταν αρκετά. Πρώτα απ' όλα ότι χρειάζεται ενίσχυση στον συντονισμό των τομεακών πολιτικών που συμβάλλουν στην ε, υλοποίηση της στρατηγικής. Η σημερινή κατάσταση, όπως είπε ένας από τους προλαλήσαντες, δείχνει ότι οι περισσότερες δραστηριότητες έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχής ή από εκεί τουλάχιστον υπάρχουν μεγαλύτερε ε, προσδοκίες. Όμως σε πολλούς από τους εμπλεκομένους φαίνεται και μοιάζει ότι η στρατηγική θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική μόνον εφόσον επιδιώκει τη συμμετοχή συγκεκριμένων ή εύστοχων τομεακών πολιτικών που μπορεί να έχουν και ιδιαίτερο αντίκτυπο όπως την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, τις μεταφορές, το περιβάλλον. Εδώ υπάρχει πραγματικά ανάγκη για περισσότερο διαφανές σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης, ώστε τα δεδομένα να είναι πιο συγκρίσιμα και επίσης υπάρχει ανάγκη να είναι και πιο λειτουργική η στρατηγική συνολικά. Γι' αυτό υπάρχει μια πρόταση για θέσπιση στόχων, όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη στρατηγική για το Δούναβη. Ένα άλλο ζήτημα είναι να ενισχύσουμε το επικοινωνιακό σκέλο τη όλη στρατηγική. Θα πρέπει να προβληθεί πολύ η στρατηγική και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό. Πρέπει να ενδυναμώσουμε την ε, ανάληψη ευθυνών και την αίσθηση του, της ιδιοκτησίας για τις διαδικασίες αυτές. Επίσης, πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των ε, βασικών εμπλεκομένων, τους συντονιστές των περιοχών προτεραιότητας, τα σημεία επαφής, τα εθνικά σημεία επαφής, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους υπευθύνους της. Τι είδους λοιπόν εργασίες προβλέπουμε για να ολοκληρώσω. Θα υποβάλουμε κείμενο με συστάσεις βασιζόμενοι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με κάποιες προτάσεις για το πώς να βελτιωθεί η στρατηγική. Στόχο μα θα είναι να διαπραγματευτούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε, στο σχηματισμό της ομάδας φίλων της Προεδρίας. Ελπίζουμε ότι θα αποσπάσουμε συμφωνία επί του κειμένου αυτού στο δεύτερο μισό του Νοέμβρη και ότι θα το εγκρίνουμε στο Γενικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο μάλλον Γενικών Υποθέσεων. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, ελπίζουμε ότι οι Δανείοι συνάδελφοι που ακολουθούν ε, στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από μας, θα αναλάβουν τη σκητάλη και θα φροντίσουν να προωθήσουν επιπλέον το θέμα αυτό, ώστε να υλοποιηθούν οι συστάσεις μας και να δημιουργήσουν ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε να ανανεωθεί απαρκώ η στατηγική σύμφωνα και με τους δεσμευτικούς στόχου που ήδη προβλέπονται στα σχετικά έγγραφα. Ευχαριστούμε κυρία Χέλντ. Τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπιτζίτσκα η οποία είναι βασική επιθεωρητής, επικεφαλής επιθεωρητής για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Σας ευχαριστώ. Η Πολωνία, όπως ακούσατε, είναι μία από τις χώρες που κατεξοχήν βρέχονται από τη Βαλτική θάλασσα και θα ήθελα για αυτό το λόγο να πω ευθύ εξ αρχή ότι αυτή η στατική για τη Βαλτική είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία που θα μας επιτρέψει να βεβαιωθούμε για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπουν και οι κανόνες της HELCOM, της Επιτροπής του Ελσίνκη. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να μιλήσω για το πρόγραμμα δράσης και τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητε της HELCOM. Η πρώτη πρωτοβουλία που η Πολωνία σκοπεύει να προωθήσει είναι η δράση η δράση μας για τις ε, χωματερές των ε, αστικών κέντρων. Εδώ χρειαζόμαστε βελτίωση των σχετικών προγραμμάτων. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας πρέπει να εξυγχρονιστούν. Απαιτούνται οικονομικές επενδύσεις μεγαλύτερες από ό,τι έχουμε ως σήμερα μόνο για το 2008 με 2009 είχαμε 4 δις σλότη ε, επενδύσεις εδώ. Σε ό,τι αφορά τις οικολογικές και γεωργικές ε, επιπτώσεις από όλη αυτή την προσπάθεια θα πρέπει θα πρέπει λοιπόν να ε, συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές εντός ενός επαρκούς ε, περιβαλλοντικού πλαισίου. Χρειάζεται περαιτέρω μείωση κατά 20% ως το τέλος του 2014 η Πολωνία θα προβλέψει και θα υλοποιήσει τις συστάσεις της Helcom για τα χημικά συστατικά. Θέλουμε να υλοποιηθούν από όλες τις χώρες της Helcom οι συστάσεις αυτές και να προστατεύσουμε έτσι και τις περιοχές της Natura 2000, αυτές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, στην ακτογραμμή το σύνολο της παράκτειας, της ακτογραμμής της Βαλτικής θα πρέπει να τη χάνει τις ίδιες μεταχείρισεις με τις προστατευμένες περιοχές. Η συμβολή της Πολωνίας στα ποσοστά φωσφόρου και αζότου που, που απορρέουν στην Βαλτική θάλασσα είναι Πολύ σημαντικά. Είμαστε τρίτοι στον φόσφορο και πέμπτη στο άζωτο. Ενώ κατά κεφαλήν τα ποσοστά των δύο αυτών χημικών ουσιών φέρνουν την Πολωνία σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα ρήπανσης για την όλη περιφέρεια. Παρόλα αυτά, παρά τους θετικούς αυτούς δείκτες, που είναι χαμηλοί ως προς τα κεφαλήν ποσοστά, καταλαβαίνουμε ότι στην Πολωνία υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος για το οικοσύστημα της ε, Βαλτικής. Όλες οι δραστηριότητε που σας παρουσίασα δεν θα είχαν υλοποιηθεί εάν δεν είχαμε λάβει κάποιους πόρους από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Επίσης, έχουμε λάβει τεχνική υποστήριξη για τους συντονιστές αυτών των ε, προγραμμάτων. Μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και σκανδιναβικά ιδρύματα που έχουν προσφέρει κονδύλια για αυτές τις πρωτοβουλίες και υπάρχουν ε, και επιπλέον πόρια από διάφορα κοινωτικά προγράμματα. Όλες αυτές τις δραστηριότητε και τα σχέδια υλοποιούνται ήδη και θα υλοποιούνται βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Θέλουμε να δημιουργηθούν σχέσει συνεργασία που να προκύπτουν από την οδηγία, τη στρατηγική και το πρόγραμμα δράση για την ευρύτερη περιφέρεια τη Βαλτική συνθήκες ε, του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ε, Βαλτική θα εξαρτηθούν από τη, τα αποτελέσματα των εμβληματικών πρωτοβουλειών σε αυτή την περιοχή. Και σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού, των θαλάσσιων υδάτων, θα χρειαστεί εδώ συνεργασία μεταξύ των κρατών τη ευρύτερη περιοχή. Χρειάζεται μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση, μεγαλύτερη ενεργοποίηση και από την Προεδρία αυτή και από τι μελλοντικέ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπιτζίτσκα. Τώρα να περάσουμε στην παρουσίαση του κυρίου Σουίτ, ο οποίος εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και εκ μέρου τη Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική, θέλω να πω εκ μέρου τη Επιτροπή Επιτροπής επίση ότι χαίρομαι πάρα πολύ που οργανώσατε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και σημαντική ακρόαση. Αρχικά, σκόπευα να σας δώσω μια γενική εισαγωγή πριν από τους ειδικού εισηγητές σας. Τώρα βέβαια ξεκίνησαν εκείνοι, οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θα έχετε ακούσει και άλλα θέματα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα. Πάντως, βάσει των συμπερασμάτων του Συμβουλίου θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά από τα προβλήματα της Βαλτικής Θάλασσας. Όπω λένε εκεί οι συνάδελφοί σα είδε από το 2006 στη διακοινοβουλευτική ομάδα για την Βαλτική θάλασσα και όλοι οι πυρογνώμονες που προσκαλήθηκαν εκεί, το συμπέρασμα ήταν ότι δεν χρειάζεται ένα νέο περιβαλλοντικό σχέδιο, αλλά μία ολοκληρωμένη και συντονισμένη στρατηγική για ολόκληρη την περιοχή. Οι τέσσερι πυλώνες λοιπόν για υφοροπεριβάλλον, για ε, ευημερούσες περιοχές, ε, για προσβασιμότητα, για ελκυστικές περιφέρειες, Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι τέσσερις πυλώνες πρέπει μεταξύ τους να είναι αλληλένδετοι για να σταθεί και να λειτουργήσει η στρατηγική για τη Βαλτική. Πρέπει να δείξουμε στους ενδιαφερόμενους, στους πολίτες των χωρών αυτών ότι η συνεργασία για όλες τις προτεραιότητες είναι η καλύτερη λύση για να τεπιστούν οι προκλήσεις και να αποφεληθούμε από τις ευκαιρίες που μας δίνει η περιοχή εκεί. Εμείς στην Επιτροπή πάντως εξεπλάγημαν πάρα πολύ από τις θετικές αντιδράσεις των πολιτών και από τον ενθουσιασμό που διαπιστώσαμε. Είδαμε ότι υπάρχει στήριξη από κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, από πρωθυπουργού μέχρι και από κοινοβουλευτικού, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, απλούς πολίτες. Στο Ταλίν πέρυσι, για παράδειγμα, είχαμε 550 νομίζω συμμετέχοντα στο πρώτο ετήσιο φόρου για την στρατηγική της Βαλτικής. Και τον Οκτώβριο στο Κτάνσκ φαντάζομαι θα έχουμε ακόμα περισσότερου. Ο ενθουσιασμό βέβαια από μόνο του δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε και δράση. Να περάσουμε δηλαδή από τα λόγια στην πράξη. Όπω ακούσατε θα έχουμε αυτή τη βδομάδα, αύριο μάλιστα, τη δημοσίευση τη πρώτη έκθεσή μα, από την οποία θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλέ δράσει. Πολλά πράγματα συμβαίνουν σε ολόκληρο το φάσμα της στρατηγικής και σε ολόκληρο το φάσμα των ε, χωρών της περιοχής, της Βαλτικής. Για παράδειγμα, για το περιβάλλον. Έχουμε προγράμματα όσον αφορά τα ναυπηγεία. Θα ακούσετε περισσότερα βέβαια από τους συναδέρφους, αλλά για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα ναυπηγεία. Επίσης για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ακούσαμε ότι η Πολωνία κάνει πάρα πολλά. Και ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω στα πλαίσια της σημερινής μας ακρόασης και κάποια άλλα προγράμματα τα οποία έχουν σαν στόχο να ε, μεταφέρουν ακόμα ε, ευρύτερα τις πολιτικές υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, είτε πρόκειται για την κοινοτροφία, είτε πρόκειται για την γεωργία κτλ. Να μην είμαστε απομονωμένοι δηλαδή, αλλά να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ αγροτών, να συμβρίσκονται, να ανταλλάσσουν ιδέες, ώστε να καταλήξουμε σε μια περισσότερο βιώσιμη γεωργία, μια περισσότερο βιώσιμη θάλασσα και επιπλέον χαμηλότερο κόστος για τους αγρότες. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ευχαριστήσουμε την HealthCom, ε, την Γενική Διεύθυνση δηλαδή, ε, αυτή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πρωτοβουλίες της στην περιοχή. βασιζόμαστε σε προτεραιότητες που έχει εντοπίσει η ίδια η HealthCom. Και όπως προχωράμε στην ανάπτυξη των στόχων μας, θα βασιστούμε στη δουλειά που έχει κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό μέχρι τώρα η ίδια η Health.com. Συνεπώς, τώρα ας δούμε ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές για την ανάπτυξη της στρατηγικής μας και την εφαρμογή της. Αποτελεί ένα μέσο offices. Αρχίζουμε να βλέπουμε τους πρώτους καρπούς των προγραμμάτων μας στην περιοχή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και το είπαν κι άλλοι, πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε ένα συστηματικό στόχο. Να ξέρουμε δηλαδή πού βαδίζουμε και ανάλογα με αυτό να αξιολογούμε τις δράσεις μας κάθε τόσο. Γι' αυτό και υπάρχει μια task force όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα κράτη-μέλη και συντονιστές από την περιοχή ώστε να αξιολογούν στους 15 χώρους στρατηγικής μας τι πρόοδος έχει επιτευχθεί. Η Task Force αυτή, λοιπόν, τέλη Σεπτεμβρίου θα πρέπει να ετοιμάσει στόχους που να λαμβάνουν υπόψη το τι δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα και να προχωρήσουμε με συνένεση πολύ περισσότερο από ότι με νομοθετικές διατάξεις. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα κάνει τη διαφορά. Για να απαντήσω στην παρατήρηση που έγινε πριν από τον κύριο Τσάρκ, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με την έκθεσή του και με τις συμβουλές του. Υπογραμμίζω λοιπόν ότι ακριβώς επειδή έχουμε όχι περισσότερα χρήματα και όχι περισσότερη νομοθεσία. Είναι τα διαφορετικά όχι τα οποία μας έχουν φτάσει, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε 50 δις για την πολιτική συνοχής υπέρ της ε, περιοχής της στρατηγικής μας. Όμως πολλά από τα χρήματα αυτά έχουν ήδη διατεθεί. Εξακολουθούμε όμως να δουλεύουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε και άλλο στην περιοχή. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει προκειμένου άλλα χρήματα και άλλες γραμμές, περιβάλλον, μεταφορές, επιχειρήσεις, καινοτομία, έρευνα, όλοι αυτοί οι τομείς να οδηγήσουν σε πολιτικές υπέρ ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που να βοηθήσει και την Βαλτική. Να υπάρχει δηλαδή περισσότερη συνοχή και μεγαλύτερο συντονισμός. Πολλά μένει να γίνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει, διευκολύνει, άντε δίνει και όθηση. Αλλά το στοιχείο κλειδί για μας είναι ότι όσοι ενδιαφερόμενοι στην περιοχή ευθυγραμμίζουν τους στόχους τους με την στρατηγική, πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρουμε υπέρ μιας πιο καθαρής βαλτικής θάλασσας και θα έχουμε κάνει τη θεωρία πράξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Ο κύριος τώρα Μαξιμίλιαν Στρότμαν που εκπροσωπεί τον Επιτρόπο κ. Σιμ Κάλλας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και από τη δική μας πλευρά. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ζητήθηκε και από τις μεταφορές να προσέλθουν, να συζητήσουν εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μας που νομίζουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει και σύγκρουση. Δηλαδή, οι μεταφορέ είναι πραγματικά θεμελιώδου σημασία για τι κοινωνίε μα, τι οικονομίε μα και πολλοί από του άλλου αγορητέ ήδη αναφέρθηκαν στην μεγάλη σημασία των μεταφορών και βεβαίω στην Βαλτική και για την σύνδεση όλων των χωρών που βρέχονται από αυτήν. Μου ζητήσατε να εξετάσω ένα θέμα μαζί σας και είναι η επερχόμενη οδηγία περιθείου. Όπως είπα, οι μεταφορές είναι κάτι που συνδέει ανθρώπους. Δεν θέλουμε να μειωθούν οι μεταφορές ούτε να παρεμποδιστούν. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά στο γεγονός ότι οι μεταφορές έχουν και αρνητικές επιπτώσεις και με τις ε, δομές τους και με τις ε, εκπομπές τους είναι γνωστά, γνωστές οι εχμές που παρουσιάζονται και σε πόλεις και αλλού και θεωρούμε ότι η ναύση πλοία, δηλαδή μετα, οι ναυτικές μεταφορές ε, προσφέρουν πλεονεκτήματα και θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν. Ιδιαίτερα αυτό ενδιαφέρει την Βαλτική και όπως είπε προηγουμένως ο Ντέιβιντ θεωρούμε πράγματι και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που οι μεταφορές έχουν ε, ενταχθεί στα δίκαια αυτή. Εδώ βέβαια είναι και τα αρνητικά. Και εδώ είναι οι εκπομπέ αερίων και θείου. Η Βαλτική, η Βόρεια Θάλασσα, υποβάλλονται σε ελέγχους σχετικά με, την, με τις εκπομπές θείου και ιδίως από τα πλοία τα οποία είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν ε, πετρέλαιο με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Το 2008 η Διεθνής Ναυτική Οργάνωση η International Maritime Organization αποφάσισε να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες λόγω του μεγάλου κινδύνου που προέρχεται από το θείο. Γιατί για την ώρα τα πλοία και είναι στην ουσία τα απόβλητα των δηληστηρίων. Αλλού ε, χρησιμοποιούνται άλλα καύσιμα, αλλά σε περιπτώσεις όπως αυτή της Βαλτικής θάλασσας οφείλουν να καταναλώνονται ε, καύσιμα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο με σημαντικά πλεονεκτήματα και για την υγεία, μείωση δηλαδή του κόστους ε, για την υγεία και ούτω καθεξής. Και ο Αμερικανός εκπρόσωπος που συναντήσαμε πρόσφατα στην Νορβηγία είπε ότι θεωρεί ότι το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθορίσει και τις δύο ακτές τους περιφέρειες ελέγχου των εκπομπών θείου θα βοηθήσει να σωθούν 6.000 ζωές τον χρόνο ο Επίτροπος Αρμόδιος για τις Μεταφορές βεβαίως μας λέει ότι όλα αυτά έχουν και ένα κόστος. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι 60 έως 80% αύξηση κόστους καυσίμων αναπλείων για την ναυτιπλοεία. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος αντικτύπων, αντίθετων δηλαδή ε, εξελίξεων, γιατί εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε να μεταφερθούν, να, ε, ε, να περάσουν οι μεταφορές από τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα περισσότερο στα πλοία. Όμως, λόγω της αύξησης του, κόστου, του κόστους, ενδέχεται το τα φορτία να μεταφερθούν ξανά, οι μεταφορές δηλαδή φορτίων, να περάσουν ξανά στους δρόμους, στις ε, οδικές μεταφορές. Οι πλειοκτήτες δεν θα σας το κρύψω και η κυρία Χάση αλλά και η Ζωάνα εδώ δεξιά μου ήταν παρούσες σε διάσκεψη με τους πλειοκτήτες οι οποίοι ανησυχούν πολύ και μας είπαν ότι ίσως υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κοινωνικές και οικονομικές, ίσως μάλιστα και περιβαλλοντικές. Ενώπιον του διλήμματος αυτού, στην Ευρωπαϊκή τουλάχιστον Επιτροπή, ο κύριος Ποτότσνικ του περιβάλλοντος και ο κύριος Κάλλας των μεταφορών συνεργάζονται χέρι με χέρι για να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες της Ένωσης, διότι αυτό που έχουμε τώρα είναι ξεκάθαρες προδιαγραφές παγκόσμια για όλες τις χώρες μέλη, αλλά και για όλα τα σκάφη που κινούνται στη Βαλτική, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να, το, να, φτιάξουμε από αυτό ένα μηχανισμό που θα κάνει πιο επίκαιρη την νομοθεσία αυτή για την προστασία από το θείο και να γίνει και δυνατόν να επιβληθεί. Και ελπίζουμε αυτό να γίνει πριν από τις θερινές διακοπές. Εμείς θα παρακολουθήσουμε αυτή την επικαιροποίηση της ε, οδηγίας ε, για να φτάσει στις ε, παγκόσμιες προδιαγραφές με ένα toolbox, ένα set μηχανισμών δηλαδή που θα λένε ή θα αγοράζει κανείς πολύ ακριβό καύσιμο χαμηλό σε θείο, χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, ή θα συνεχίζει να καταναλώνει το ε, φθηνό καύσιμο που είναι υψηλής περιεκτικότητα σε θείο, αλλά θα καθαρίζει εκ των υστέρων τα καυσαέρια με ε, συσκευές που λέγονται στα αγγλικά scrubbers. Εμείς θεωρούμε ότι το καλύτερο είναι το LNG, το αέριο δηλαδή που είναι πολύ ε, καλύτερο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι για την ώρα δεν έχουμε ούτε σκάφη, ούτε η απαραίτητη υποδομή. Άρα είναι, το θέμα αρχαίως είναι πρώτο σηκώτε τα αυγό. Αλλά τώρα αυτό που θα χρειαστεί είναι να φτιάξουμε ένα δίκτυο αποθηκών του LNG. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε σημαντικές επενδύσεις, να βοηθήσουμε και τα κράτη αλλά και την ε, βιομηχανία να επενδύσουν σε νέα τεχνολογία η οποία θα προσφέρει μια στέρεα βάση για τη μελλοντική εξέλιξη της ναυσιπλοείας αλλά και ειδικότερα βέβαια ε, των χωρών που βρέχονται από τη Βαλτική θάλασσα. Ευχαριστούμε κύριε Στρότμαν. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της ακρόασής μας, εκτός και αν υπάρχουν ερωτήσεις. Θέλει κάποιος να θέσει ερωτήσει στου συμμετέχοντε αυτό το πάνελ. Ωραία. Περνάμε στο δεύτερο μέρος λοιπόν. Ε, Βαλτική θάλασσα, η πλέον ε, μολυσμένη θάλασσα παγκοσμίω. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Προσκαλώ τον κύριο Μίκαελ Ντούρκιν, Ντέρκιν, μέλος της ε, Γραμματείας της Επιτροπής του Ελσίνκη για την προστασία της Βαλτικής θάλασσας. Σας προσκαλούμε εδώ στο βήμα. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας και ψηφιστικής ασφάλειας και περιβάλλοντος που μας προσκάλεσε να μιλήσουμε εδώ για, το, περιβαλλοντικά, περιβαλλοντικά θέματα της Βαλτικής θάλασσας. Να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους ε, του, της γραμματέως της Επιτροπής. Δεν ήταν εδώ λόγω ελλημένων υποχρεώσεων Συναντήσει δηλαδή με κάποιου από τους ε, συνεργάτες μας να είναι εδώ μαζί σα. Στην παρουσίασή μου, αν θέλετε περάσετε στην επόμενη διαφάνεια, θα προσπαθήσω να περιγράψω σύντομα, παρόλο που δεν είναι απλό εγχείρημα, τι πρέπει να κάνουμε για να θεραπεύσουμε τη Βαλτική θάλασσα. Και θα αφιερώσω και λίγο χρόνο σε μερικές διαφάνειες εξηγώντα ποιο είναι το νόημα για μα τη Βαλτική θάλασσα, τι είναι η HELCOM συνοπτικά και ποια είναι πολιτική, το πολιτικό πλαίσιο τη HELCOM σε ό,τι αφορά την ανάκτηση και την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής. Για να ξεκινήσω να σας δώσω το γενικότερο πλαίσιο. Η Βαλτική θάλασσα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος ε, των, ε, της συνολικής επιφάνειας των ωκεανών. Περίπου 10 έως 15% των παγκόσμιων μεταφορών επίσης. Όλα αυτά στα πλαίσια μιας θάλασσας που είναι ευαίσθητη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών ενώ η ανανέωση των υδάτων είναι πολύ χαμηλή, το ποσοστό ανανέωση είναι πολύ χαμηλό. Ό,τι μπει στη Βαλτική θάλασσα ε, μένει για περίπου 30 χρόνια, ενώ είναι υφάλμηρο το νερό, δηλαδή θαλάσσια και είδη υλικών υδάτων συγκατοικούν. Ω προ τι μεταφορέ, η θαλάσσια περιοχή τη Βαλτική ε, επηρεάζεται από τον ευτροφισμό. Ευτροφισμό με διπλάσια ε, αύξηση στην περιεκτικότητα σε τέτοιε ουσίε τον τελευταίο αιώνα. Επίση, αυτό το ποσοστό είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι στο βορειοανατολικό Ατλαντικό, λόγου χάρη. Δεν θα πρέπει όμω να ξεχνούμε. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η ξεκάθαρη οικονομική αξία που παράγει η βαλτική για τους ε, ε, ανθρώπους που κατοικούν παρακτίως της θάλασσας είναι 5 δις ευρώ ετησίως. Ακούμε ότι πολλές ανθρωπογενείς δραστηριότητες καταστρέφουν το περιβάλλον της Βαλτικής. Τα περιδάγματα περιλαμβάνουν τις μεγάλες απορροές ε, γεωργικών πεσμάτων ε, στην ε, Βαλτική, την τα αστικά λίμματα στην Ανατολική, ιδίω Βαλτική, και αυτό δυσκολεύει και όσου εργάζονται και όσου κατοικούν και ακόμη γίνεται αδυνατό να κολυμπήσει κανεί. Επίση, ε, υπάρχουν είδη τα οποία κανονικά χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση όταν αλλιεύονται και τα οποία οδεύουν προ την ε, εξαφάνισή του. Μιλήσαμε για την υψηλή συγκέντρωση διοξίνη σε ψάρια το ε, πρωί. Σύμφωνα με του ευρωπαϊκού κανονισμού, τα ψάρια που αλλιεύονται στην Βαλτική δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται. Επίση, γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Έχουμε πολύ έντονες πτήσεις, ε, πτήση αεροπορικό πάνω από, πτήσεις αεροπλάνο πάνω την Παλτική και επίσης ιδιαίτερες καιρικέ συνθήκες. Όλα αυτά επηρεάζουν ε, τις συνθήκε. συνθήκες. Να σας παρουσιάσω τώρα την ε, οργάνωση την οποία προέρχομαι. Η Helcom είναι μια επιτροπή από εννέα ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής ε, και την ε, καταπολέμηση της ρήπανση καθώς και τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοείας. Είμαστε το κυβερνών ε, σώμα για την ευρύτερη διασφάλιση της περιοχής της Βαλτικής που είναι γνωστή ως Σύμβαση του Ελσίνκη αυτή η σύμβαση υπογράφηκε από όλα αυτά τα κράτη το 1974 ε, και ανανεώθηκε το 1982 ε, από τι πολιτικέ εξελίξει στην ευρύτερη περιοχή. Βασιζόμαστε στη συνεργασία μεταξύ των χωρών τη Βαλτική και τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ώστε να μπορέσουμε να καταρτήσουμε συγκεκριμένε πολιτικέ για την περιοχή τη Βαλτική. Από το 2010 πρέπει να τονίσουμε ότι η Χέλκομ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο για το συντονισμό πλατφόρμα για την περιφερειακή υλοποίηση τη Ευρωπαϊκή Θαλάσσια ε, και στρατηγική για την Βαλτική. Όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και αδυναμίε, όχι μόνο δυνατά σημεία για την Επιτροπή μας και υπάρχουν και προβλήματα δυσεπίλητα. Για το λόγο αυτό η υπουργική συνάντηση τη Χέλκομ το 2007 στην Κρακοβία υιοθέτησε ένα πρόγραμμα δράση το οποίο ήδη αναφέρθηκε. Το πρόγραμμα αυτό δράση άνοιξε το δρόμο για το να αναλυφθεί δράση και μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντο. Το πρόγραμμα δράση υιοθετεί μια προσέγγιση για την προστασία των οικοσυστημάτων σε σχέση με τι ανθρωπογενεί δραστηριότητε και επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα ευτροφισμό, επικίνδυνε ουσίε, θαλάσσιε δραστηριότητε φιλικέ προ το περιβάλλον και προστασία τη βιοπικιλότητα. Επιπλέον, οι έννοιε και οι προσεγγίσει τη Χέλκομ χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλε διεθνεί προσεγγίσει, όπω την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και την Προστασία τη Βαλτική. Με μεγάλη χαρά ακούσαμε ότι η στρατηγική αυτή θα προωθηθεί περαιτέρω με δείκτε ε, και στοιχεία και την πείρα που ήδη διαθέτουμε στη Χέλκομ. Όλα αυτά έχουν ενισχύσει τι σχέσει συνεργασία και τη δυνατότητα ενσωμάτωση πολιτικών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντο τη Βαλτική. Θα βρείτε περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα δράση στον ιστότοπο μα. Ωστόσο, για να απαντήσω στην ερώτηση του πώ θα θεραπευτεί η Βαλτική, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ποια είναι η κατάσταση υγεία του ασθενού για τον οποίο συζητούμε. Αυτή ήταν και η βάση για το πρόγραμμα δράση ε, τη Βαλτική όταν άρχισαμε να εργαζόμαστε. Μια σφαιρική αποτίμηση τη υγεία των οικοσυστημάτων στη Βαλτική. Πράγμα που έγινε λίγο καθυστερημένα βέβαια σε σχέση με την υιοθέτηση του προγράμματο δράση τη Βαλτική. Η αρχική αξιολόγηση δείχνει μια σφαιρική παρουσίαση τη θαλάσσιου περιβάλλοντο το 2003 και 2007 και τι ενδιάμεσε εξελίξει. Βλέπουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν εργαλεία θεματικών αξιολογήσεων και καταμέτρησης της κατάστασης για να δούμε την υγεία του οικοσυστήματος στην Παλαιτική. Οι εκθέσεις της προσέγγισης αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω σημεία αναφορά γιατί προηγήθηκαν του προγράμματο δράση για την Βαλτική. Εάν θέλουμε να δούμε κατά πόσον τα μέτρα που αναλύθηκαν βελτίωσαν την κατάσταση υγεία τη Βαλτική. Η αρχική ολιστική αυτή προσέγγιση ασχολείται ακριβώ και με την κατάσταση υγεία των οικοσυστημάτων και τι πιέσει που δέχεται ανθρωπογενώ στο θαλάσσιο περιβάλλον. Φαίνεται από την αξιολόγηση ότι η υγεία είναι πολύ κακή για, την, για το σύνολο τη Βαλτική. Βλέπετε ότι οι περιοχέ που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα υγεία έχουν ε, κόκκινο χρώμα, ενώ αυτέ που έχουν μικρότερο κίτρινο. Οι ανθρωπογενεί δραστηριότητε ασκούν πίεση στο σύνολο τη ε, περιοχή. Το βλέπετε με, με πορτοκαλί ε, κόκκινο και κίτρινο τις περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα. Εκεί όπου υπάρχουν λιγότερα προβλήματα, το χρώμα είναι διαφορετικό όπως τον κόλπο της ε, Βοτνίας. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι ο αντίκτυπος είναι σοβαρός από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η ρήπανση ε, αφορά κυρίως τα ανοιχτά ύδατα της, αλφί της Βαλτικής, αν και τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζονται στις παράκτιες, στις πιο ευαίσθητες περιοχές στις ανοιχτέ λεκάνες τα προβλήματα προέρχονται από αλλιευτικέ δραστηριότητε, καθώς και την ατμοσφαιρική εναπόθεση επικίνδυνων ουσιών ενώ υπάρχει και ο ευτροφισμός ως πρόβλημα που επηρεάζει την βιοπικιλότητα και την καλή κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων από που δεν μπορούν πλέον να αποσπαστούν υπηρεσίε. Η οικονομική ανάλυση που συμπεριλαμβάνεται στην ολιστική προσέγγιση είναι... Ε, δείχνει ότι είναι δαπανηρέ οποιασδήποτε προσπάθειε αποκατάσταση, αλλά αν δεν αναλάβουμε καμία δράση, το κόστο θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Για τη διαδικασία τώρα υλοποίηση του προγράμματο δράση για την Παλτική. Ξέρουμε ότι ένα πράγμα είναι να συμφωνεί κανεί στο διεθνέ επίπεδο τι πρέπει να γίνει, αλλά προκειμένου όλα αυτά να υλοποιηθούν και να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο τα μέτρα. Γι' αυτό το πρόγραμμα δράση τη ΧΕΛΚΟΜ δηλώνει ότι όλε οι χώρε πρέπει να ορίσουν εθνικά προγράμματα δράση, συγκεκριμένα για τον ευτροφισμό και τι επικίνδυνε ουσίε. Ένα χρόνο μετά την Υπουργική Σύνοδο στην ε, Μόσχα πέρσι, ε, όπου έγινε και αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων δράση, ε, βρίσκουμε καλά παραδείγματα, αλλά και περιοχέ όπου χρειάζεται περαιτέρω στήριξη. Το επόμενο στάδιο θα είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των αναλυθέντων μέτρων και να δούμε αν επιτέχθηκαν οι στόχοι που είχαν ε, τεθεί και αν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα. Θα πρέπει εδώ να αποφεληθούμε και από τα ευρωπαϊκά πλαίσια και προγράμματα, όπως την οδηγία για την ποιότητα των ε, αστικών, ε, για την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων και την προστασία του θαλάσσιου, του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ένα από τα πιο επίγοντα προβλήματα της Βαλτικής είναι ο αστροφισμός. Εδώ πρέπει να προβλεφθούν μέτρα προκειμένου να υπάρξει καλύτερη υγεία στο νερό της Βαλτικής ό,τι αφορά τον ανθρωπισμό, στο 2016. Θα σας αναφέρω μόνο μερικά καλά παραδείγματα όσων αξιολογήθηκαν από τα εθνικά προγράμματα δράσης καθώς και για τις εξελισσόμενες δραστηριότητε μετά την έγκριση του προγράμματος δράσης για την Βαλτική. Μερικά από αυτά ήρθαν εις πέρα και με την οικονομική στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαμβάνονται λοιπόν οι μεγάλε ε, Τη της Πολωνίας για την διαχείριση και την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, αλλά εδώ και η Αγία Πετρούπολη και η Ρήγα και η Σρέτσιν και άλλε πόλει ε, παράκτια της Βαλτικής ή του εσωτερικού εσωτερικούς ε, υδάτινους δρόμους έχουν αναλάβει μέτρα. Κάποιες φορές πρέπει να είναι πιο αυστηρά τα μέτρα και από την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, όπως με το πρόγραμμα PURE τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε περήφανοι επίση για του εθνικού κανόνες ε, για την ε, εξάλληψη του φωσφόρου από τα οικιακά απορριπαντικά που έχουν αναλυφθεί στη Σουηδία, τη Λετωνία και η Φινλανδία, καθώς και η Γερμανία προγραμματίζουν να αναλάβουν σχετικά μέτρα. Περιμένουμε όμως να δούμε και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θέμα αυτό. Υπάρχουν επίσης ε, νέοι κανόνες για την απορροή λιμάτων από τα επιβατικά σκάφη και ειδικέ περιοχέ όπω ορίζονται από τη σύμβαση Μάρπολ. Εδώ ε, χρειάζονται όμω ειδικέ εγκαταστάσει στου λιμένε ε, για τα μεγαλύτερα λιμάνια που υποδέχονται επιβάτε και αυτά πρέπει να προβλεφθούν το αργότερο στο 2015. Αυτό το μελετούμε με τουλάχιστον πέντε μεγάλε πόλει λιμένε στην ε, Βαλτική. Πρέπει επίση να δούμε ποιε είναι οι πηγέ και ποιοι οι δρόμοι που ακολουθούν συνήθω οι επικίνδυνε ουσίε στη Βαλτική. Εδώ υπάρχει ήδη πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκής, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοχύμπα και πέραν ε, του ευτροφισμού και των επικίνδυνων ουσιών έχουμε και άλλα προβλήματα όπως τα λίματα και η θαλάσσια κίνδυνη. Δεν θα πρέπει εδώ να ξεχάσουμε ότι πέραν των πανευρωπαϊκών προγραμμάτων και σχεδίων στα οποία συμμετέχουμε, συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη που είναι γειτονές μας ε, στους ε, υδάτινους αυτούς πόρους της Βαλτική. όπως η Ρωσία που επηρεάζει την Βαλτική με την Αγία Πετρούπολη και το Καλίνιγκρατ. Δεν θα σταθώ στις επόμενες διαφάνειες, θα έλεγα να περάσουμε κατευθείαν σε συμπεράσματα. Διότι μπορείτε να τα δείτε στο αντίτυπό σας στα σημεία που έχω αναφέρει και ποιε θεωρώ ότι είναι σημαντικότερε δράσει, όπω και πού χρειαζόμαστε περαιτέρω στήριξη. Για να συμπεράνω, η διευκόλυνση χρήση ε, στοχευμένων λύσεων για την πολιτική είναι σημαντική με περιφερειακή προσέγγιση. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε λύσει που να καλύπτουν την, ε, τον ευαίσθητο χαρακτήρα τη Βαλτική. Χρειάζεται πολιτική δέσμευση, αν και ήδη έχει αναλυφθεί κάποια δράση, για να στηριχθεί ε, το πρόγραμμα δράση για την πολιτική. Από τα ανώτερα πολιτικά επίπεδα και ήδη από τη Σύνοδο για την Βαλτική που έγινε το Φεβρουάριο του 2010 φάνηκε αυτό. Εκεί συμμετείχαν αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων. Ε, Επίση, χρειάζεται Διάλογο με του ενδιαφερομένους. Ακούσαμε στους προηγούμενους ε, λόγους να αναφέρεται αυτό και ο διάλογος αυτός πρέπει να ενισχυθεί και στα πλαίσια της Χέλκομ ε, προβλέποντας νέα φόρα με τις συζήτηση με τι γεωργικέ αρχέ, τι αρχέ υπεύθυνε για την αλληλεία, το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει ευκαιρίε για τέτοιο διατομεακό διάλογο. Επίση, υπάρχει ανάγκη περισσότερο στοχευμένης χρηματοδότησης για συγκεκριμένα προγράμματα στην περιοχή. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη με τα νέα κονδύλια και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προκύπτουν από τα περιφερειακά προγράμματα. Και να μην ξεχνάμε και τη διασυνοριακή ρήπανση. Πέραν των παρακτήων κρατών υπάρχουν και άλλες χώρες στο υδάτινο αυτό μέτωπο που μπορεί να μην είναι ε, άμεσα συμβάλλονται στο όλο πρόβλημα, αλλά να μπορούν να αποφεληθούν από τι λύσει. Αυτό το θέμα θα είναι πολύ σημαντικό, όπω ακούσαμε, για την επερχόμενη πολιτική προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι θα ενισχύσει τι προσπάθειε για μια υγιέστερη Βαλτική θάλασσα. Σα ευχαριστώ. Και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι από το Ίδρυμα για την ε, Βαλτική και από το Φιλανδικό Ινστιτούτο θα με συμπληρώσουν στα θέματα του ευτροφισμού. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπο Γκούσταυσον, επιστήμονας στο Ινστιτούτο για τη θάλασσα, για θαλάσσια μοντέλα της Στοκχόλμης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα. Το Ινστιτούτο μας, Baltic Nest, έχει εταίρους και στη Φιλανδία και στη Δανία. Εγώ διευθύνω το σουηδικό τμήμα που χρηματοδοτείται εν μέρη από την σουηδική κυβέρνηση. Μια από κύριους στόχος του είναι να βοηθά την Helcom με επιστημονικά δεδομένα για να βοηθήσει την πολιτική διαδικασία. Έτσι λοιπόν σήμερα θα επικεντρωθώ στο πώς εμφανίζεται σήμερα η Βαλτική και πώς ήταν πριν από 100 χρόνια και πώς ελπίζουμε ότι θα είναι στο μέλλον. Να τη είχαμε πριν, τα κιανοπράσινα φύκια, τα οποία σήμερα αποτελούν μεγάλο πρόβλημα στη Βαλτική θάλασσα. Πριν από 15 χρόνια ήταν έτσι περίπου τα πράγματα και αυξάνονται κάθε χρόνο στη Βαλτική. Και αν υπολογίσουμε την αύξηση αυτή, είναι 9 φορές παραπάνω από ό,τι τον προηγούμενο αιώνα. Το ίδιο και με την παραγωγή ε, γενικότερα. Έχουν πολλαπλασιαστεί επί τρία. Κάτι το οποίο οδηγεί και σε αυτό το ειδικό φύκι στις ακτές και μειώνεται έτσι η ορατότητα, κάτι το οποίο επηρεάζει και την αλίευση. Μια επιπλέον συνέπεια της αύξησης των φυκιών είναι ότι βυθίζονται, ε, πάνε στο βυθό δηλαδή κατακάθονται και απορροφούν οξυγόνο. Έτσι λοιπόν, στα βαθιά έχουμε όλο και μεγαλύτερη επέκταση επί έξι τα τελευταία χρόνια των υπόξικων δηλαδή βυθών. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι τα ειζήματα, κάτι το οποίο μπορείτε να δείτε από παλιά πώς ήταν. Και τι βλέπουμε απάνω, τη μείωση του οξυγόνου. Κάποια στιγμή βέβαια συνέβη κάτι στο ίσμα το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί. Και τώρα έχουμε καινούργια στοιχεία που μας έρχονται από διάφορα προγράμματα που δείχνουν ότι η κατάσταση στη Βαλτική σήμερα είναι μοναδική. Ποτέ δεν ήταν έτσι σε όλη της την ιστορία. Συνεπώς, γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο. Εδώ βλέπετε ένα σχέδιο. Το πράσινο δείχνει πώς οι απορροές συσσωρεύονται στην ε, Βαλτική θάλασσα και πώς εξελίσσονται αυτές. Το παράδοξο εδώ είναι ότι στις περισσότερες χώρες, σε όλες τις χώρες, ξεκινήσαμε να μειώνουμε τις απορροές αυτές εδώ και 30 χρόνια. Και η μείωση είναι σημαντική. Παρόλα αυτά βλέπετε τη μαύρη γραμμή που είναι η βιομάζα που περιλαμβάνει τα διάφορα βακτηρίδια κτλ. Αυτή αυξάνει λοιπόν συνεχώς. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν χρονικά κάποιες διακοπές. Για να καταλάβουμε και να προβλέψουμε τις επιπτώσεις, χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα που να μας περιγράφουν το ίδιο το φαινόμενο. Και αυτό κάνουμε εμείς στην Baltic Nest αναπτύσσουμε μοντέλα, προτείνουμε λύσεις βάσει μιας ολιστικής προσέγγισης για τη Βαλτική θάλασσα. Είναι ένα μοντέλο λοιπόν που χρησιμοποιούμε και εδώ, όπου προχωράμε σε μια εκτίμηση. Το άζωτο και ο φόσφορος πόσο απελευθερώνονται στα βάθη της θάλασσας και τι περιθώρια έχουν για να εξακολουθούμε να έχουμε ένα αποδεκτό περιβάλλον. Ποιο θα είναι το μέλλον τώρα. Παρόλο που τα πράγματα δείχνουν άσχημα σήμερα, θα βελτιωθούν. Και θα βελτιωθούν γιατί όπως είπαμε υπάρχουν κάποιες διακοπές στο σύστημα. Η επιδείνωση δεν συνεχίζει δηλαδή. Και αν καταφέρουμε να περιορίσουμε τις απορροές που είναι η πράσινη γραμμή που, βλέπατε, που βλέπετε εδώ, βλέπετε ότι υπάρχει μια φθήνουσα απορία της πράσινης γραμμής. Αν δηλαδή προχωρήσουμε και εφαρμόσουμε το πρόγραμμα δράσης για τη Βαλτική που αναφέρεται στις ανώτατες απορροές, αν λοιπόν καταφέρουμε και το τηρήσουμε, τότε μπορεί να καταλήξουμε στην μαύρη γραμμή που σημαίνει ότι θα συνεχίσει η κατάσταση όσο έχει τώρα ή αν τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου, ξεφύγουν από τον ελεγχό μας, τότε θα διηγηθούμε στην πορεία της μπλε γραμμής, που σημαίνει ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Εγώ πιστεύω όμως ότι οι κυβερνήσεις γύρω από την Βαλτική μπορούν να αναλάβουν μια μοναδική ευθύνη σήμερα για να αποφύγουν ε, την ευτροφία. Θα πάρει χρόνο βέβαια, αλλά μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Όμως, μια στιγμή, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο, μια επιπλοκή. Και αυτή είναι οι κλιματικές αλλαγές. Κάτι με το οποίο έχουμε αρχίσει να ασχολιόμαστε με το πρόγραμμα Bonus, όπου έχουμε ένα πρόγραμμα για την στήριξη του οικοσυστήματος όπως συμμετέχουν η Γερμανία, η Φιλανδία, η Εστονία, η Πολωνία και η Δανία. Όπου προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας όλα τα προγράμματα του IPCC και να δούμε πώς αυτά επηρεάζουν την κατάσταση στη Βαλτική θάλασσα και πώς επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα των δικών μας των μέτρων όσον αφορά την ευτροπία. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα η θέρμανση του πλανήτη θα οδηγήσει σε περισσότερη ευτροφία. Αυτό όμως Σημαίνει συγχρόνως ότι όσο περισσότερο μειωθούν ε, οι απορροές, τόσο πιο σημαντικό θα είναι αυτό. Μην το ξεχνάμε. Δηλαδή ότι αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη σημασία η μείωση των γεωργικών απορών. Συμπεράσματα. Ο λόγος που είναι η Βαλτική όπως είναι, είναι οι γεωργικές απορές όπως είπαμε, δεν είναι απελπιστική η κατάσταση, οι χώρες γύρω από τη Βαλτική έχουν ήδη αναλάβει δράση για να τις μειώσουν και λαμβάνουν ε, δράσεις και αποφάσεις για να τις μειώσουν ακόμα περισσότερο και να βελτιωθεί η κατάσταση. Θα πάρει όμως χρόνο για να έχουμε ανάκαμψη και αποκατάσταση. Οι μειώσεις πάντως στις απορροές αποκτάνε όλο και μεγαλύτερη σημασία προς τα τέλη του αιώνα, όταν η θέρμανση του πλανήτη θα επηρεάσει περισσότερο και τη Βαλτική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκούσταυσον. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σέπο Κνουτίλα από το ΣΑΙΚ που είναι το Φιλανδικό Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να προσέλθω εδώ στην Ευρωβουλή και να σας πω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βαλτική και κυρίως για Απορροές. γεωργικών ε, ε, Για, θα δείτε πρώτα εδώ αναχώρα τις γεωργικές απορροές χωρισμένες στη διαφάνεια αυτή κατά πηγή. Κοιτάξτε τα ερυθρά και πράσινα χρώματα στους κύκλους αυτούς. Τα, τα... τα ερυθρά χρώματα δείχνουν ότι προέρχονται από τοπικές κοινότητες. 80-90% είναι λοιπόν από ε, τοπικές κοινότητες. Το σκούρο πράσινο δείχνει άλλες ε, πηγές 80% περίπου από την γεωργία που καταλήγουν όπως είπα στην Βαλτική. την ε, τελευταία δεκαετία έχουμε προχωρήσει σε καθαρισμό μεγάλου ποσοστού των υδάτων που έρχονται από διάφορες τοπικές κοινότητες. Στην διαφάνεια αυτή θα δείτε την μείωση τα τελευταία 40 χρόνια σε όλες τις χώρες, κυρίως ε, του ε, φωσφόρου φωσφορικών ενώσεων που προέρχονται από τις τοπικές κοινότητες στο δεξί μέρος της διαφάνειας που είναι πάνω από 25.000 τόνους όπως είπα στη δεξιά και η κιανή γραμμή δείχνει το σημερινό φόρτο ε, φωσφόρο από όλες τις πηγές που καταλήγουν στη Βαλτική θάλασσα. Αν λοιπόν δεν είχε γίνει τίποτα την τελευταία, ε, τις τελευταίες μάλλον δεκαετίες για να μειωθεί ο φόρτος από η επιβάρυνση δηλαδή από τις τοπικές κοινότητες θα ήταν σχεδόν διπλάσια η ποσότητα που θα δεχόταν η Βαλτική θάλασσα σήμερα. Όπως είπε ο συνάδελφος Γκούσταψεν, η μείωση των απορών στις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε σημαντική, αν και δεν το βλέπουμε αυτό ε, ακόμα στην κατάσταση της Βαλτικής. Παρόλο λοιπόν που έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την μείωση των απορροών από τις τοπικές κοινότητες. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στις περισσότερες ε, χώρες που βρέχονται από τη Βαλτική θάλασσα. Έχουμε υπολογίσει το, ε, το απομένον δυναμικό φωσφόρου και αζότου για μείωση δηλαδή των ε, επιβαρύνσεων από τις τοπικές κοινωνίες και τα νούμερα αυτά δείχνουν σε όλες αυτές τις χώρες και στη Λευκορωσία παρόλο που δεν είναι ε, μέλος της ΕΛΚΟΜ συνολική, συνολικό δυναμικό μείωσης βλέπετε στην, στην ερυθρή στήλη είναι ακόμα υψηλή εάν συγκριθεί με το συνολικό φόσφορο που καταλήγει σήμερα στην Βαλτική θάλασσα μπορεί να μειωθεί ακόμα κατά 20% με μείωση των απορροών φωσφορικών ενώσεων από τις ε, διάφορες τοπικές κοινότητες. Στο σχέδιο δράσης της Helcom για τη Βαλτική συνιστάται να γίνει προσπάθεια να φτάσει στο 90% η μείωση των ε, φωσφορικών ενώσεων που απορρέουν στην ε, Βαλτική πέραν και του στόχου της ε, κοινοτικής οδηγίας που βάζει στόχο το 20%. Μέχρι το 90% λοιπόν. 10% λοιπόν της 100 παραπάνω από τις ετήσιες απορροές φωσφορικών ενώσεων. Αυτός ο στόχος Helcom είναι πολύ σημαντικός για όλες τις χώρες που ε, περικλείουν την ε, Βαλτική θάλασσα. η ίδια πληροφορία τώρα εδώ για το άζωτο. Δεν βλέπουμε να υπάρχει το ίδιο δυναμικό μείωση όπως για τον φόσφορο. Είναι σημαντικό ωστόσο να επενδύσουμε και στον τομέα αυτό διότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό ο πλευράς κόστους να μειωθεί η επιβάρυνση από άζωτο από τις κοινότητες, τοπικές κοινότητες σε σχέση για παράδειγμα με τη γεωργική παραγωγή. Στην ε, διαφάνεια αυτή θα δείτε το σύνολο της επιβάρυνσης από ενώσεις μέσω των νερών που καταλήγουν δηλαδή στην ε, Βαλτική θάλασσα με επίπεδο παρόμοιο με σήμερα. Η ερυθρά είναι η σημερινή επιβάρυνση Το maximum που, προβλέπει η Helcom είναι στην πράσινη στήλη και η επόμενη στήλη είναι πόσο θα πρέπει να μειωθεί η επιβάρυνση από φωσφορικές ενώσεις για να επιτευχθεί ο στόχος του Action Plan για τη Βαλτική με την έννοια ότι, ότι θα μπορούμε να επιτύχουμε μέχρι το 2021 μια ανεκτή κατάσταση στη Βαλτική, μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση στην Αττική με αυτό το MWWP που βλέπετε που είναι μηχανισμοί δηλαδή ε, επεξεργασίας των ε, υγρών αποβλήτων από τις ε, τοπικές κοινότητες. Και μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερη μείωση αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μειωθεί η από τη γεωργία κατά 5.000, κατά τόνους ετησίως. Το ίδιο για το άζωτο τώρα, όπως για τον φωσφόρο, ...η κύριοι τομείς όπου μπορούμε να οδηγηθούμε σε σημαντική μείωση σε υγρά απόβλητα είναι πάλι οι τοπικές κοινότητες με εγκαταστάσεις καθαρισμού που είναι ακόμα πιο σημαντικές για το άζωτο για να μειωθεί δηλαδή η επιβάρυνση από γεωργικά απόβλητα. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τόσο πολύ όπως για το φόσφορο στο επίπεδο των τοπικών κοινοτήτων. Για την ιστορία τώρα των γεωργικών αποβλήτων, πώς, πού αρχίζει και πώς έχει εξελιχθεί στις τελευταίες δεκαετίες. Σε Αυτήν την διαφάνεια βλέπετε φωσφόρο και άζωτο και συγκέντρωση στην ε, Βαλτική από το 1950 μέχρι το 2010 και θα δείτε ότι οι συγκεντρώσεις αρχίζουν να αυξάνονται και με ταχύ ρυθμό μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι έγινε τότε στον γεωργικό τομέα. Μετά από το δεύτερο πόλεμο αρχίζουν να χρησιμοποιούνται περισσότερο τα τεχνητά λοιπάσματα στις δυτικές χώρες. Βλέπετε εδώ στη διαφάνεια αυτή την παγκόσμια παραγωγή λιπασμάτων και βλέπετε πόσο απότομα αυξάνει η καμπύλη μετά από το 1945. Ο βασικός λόγος που κρύβεται πίσω από αυτή την εξέλιξη είναι ότι πριν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν κλειστό το κύκλωμα της ε, λίπανσης στη Γεωργία. Δηλαδή τα ε, απορρίμματα ε, της Γεωργίας χρησιμοποιούνταν ως λίπασμα και δεν χρησιμοποιούνταν τεχνητά λιπάσματα. Ενώ μετά έσπασε ο κύκλος αυτός και χωρίστηκε η παραγωγή, η φυτική παραγωγή και η ζωική παραγωγή. Επομένως, η κοπριά δεν χρησιμοποιούνταν πλέον ως ε, η πιο σημαντική πηγή φωσφόρου και αζότου για την παραγωγή σιτηρών. Εδώ βλέπετε στις στήλες αυτές για το άζωτο και για τον φωσφόρο που παράγονται την λεκάνη της Βαλτικής από όλες τις χώρες και από όλο τον ανθρώπινο πληθυσμό και τα τεχνητά λοιπάσματα που χρησιμοποιούνται στη λεκάνη της Βαλτικής και θα δείτε επίσης στη δεξιά στήλη άζωτο και φωσφόρο που περιλαμβάνονται στην κοπριά των ζώων που παράγεται γύρω από τη λεκάνη της Βαλτικής. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσες ε, τροφικές ύλες, ε, πόσο έχει αυξηθεί η πίεση των ε, αποβλήτων αυτών μετά από την έναρξη χρήσης τεχνητών λοιπασμάτων στη Γεωργία. Και σήμερα, επειδή η παραγωγή σιτηρών και παραγωγή, η κτηνοτροφική παραγωγή έχουν χωριστεί, όλη η κοπριά που παράγεται ετησίως στην κτηνοτροφία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα γιατί είναι τόσο συγκεντρωμένες, ε, συγκεντρωμένο το υλικό αυτό γύρω από τα αγροκτήματα που δεν είναι αρκετά ώστε να και δεν είναι αρκετά μάλλον να χρησιμοποιηθούν ώστε σε ορισμένες περιοχές η κοπριά των ζώων δεν αποτελεί παρά απόβλητο Και κάτι άλλο που επιταχύνεται με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη μάλλον, μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα τελευταία δηλαδή 50 χρόνια, η κατανάλωση κρέατος έχει αυξηθεί σημαντικά. Προ 50 ετών που καταναλώναμε το μισό περίπου, περίπου του κρέατος που καταναλώνουμε σήμερα. Όσο περισσότερο κρέας καταναλώνουμε, τόσο περισσότερες γέες χρειαζόμαστε για την εκτροφή των ζώων και στις περισσότερες δυτικές χώρες και στη Φιλανδία και στη Σουηδία 70 έως 80% των γεών χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ζωοτροφών για την κτηνοτροφία. Συμπεραίνοντας για τη γεωργία με η στόχοι μείωσης για την επιβάρυνση της Βαλτικής είναι σημαντική μεν οι αποτελούν πραγματική πρόκληση. Ταυτόχρονα μέχρι το 2050 θα αυξηθεί η ζήτηση τροφίμων παγκοσμίως τουλάχιστον κατά 50%. Ταυτόχρονα οι αλλαγές του κλίματος θα καταστήσουν πρακτικές της γεωργίας πιο ελκυστικές, ε, τουλάχιστον στο βόρειο μέρος της ε, λεκάνης της Βαλτικής, αυξανόμενες λοιπόν, αύξηση μάλλον θερμοκρασιών και παραγωγή επομένως ε, απορών θα είναι σημαντικότερη και στο μέλλον θα αυξηθούν και οι τιμές των τροφίμων και επομένως θα γίνει και οικονομικά πιο ελκυστική η γεωργική παραγωγή. Βλέποντας βέβαια αυτά εδώ είναι δύσκολο να πιστεύσει κανείς ότι θα μειωθεί, θα μειωθεί η, παραγωγή, η γεωργική παραγωγή γύρω από την λεκάνη της Βαλτικής. Αυτό που ενδιαφέρει πάντως είναι να μειωθούν οι πηγές φωσφόρου και για το μέλλον για να μπορεί να ασκείται η γεωργία οπουδήποτε ανά τον κόσμο η προϋπόθεση θα είναι οπωσδήποτε ανακύκλωση, ανακύκλωση του φωσφόρου με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό βέβαια θα οδηγήσει τελικά σε μείωση των απορών φωσφόρου στη Βαλτική θάλασσα. E, Ευχαριστούμε κύριε Κνουτίλα για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Μακάρι να μπορούσαμε να φανταστούμε γεωργία που να χρησιμοποιεί λιγότερα λιπάσματα με περιεκτικότητα σε άζωτο. Θα ήταν πολύ ωραία να επιστρέψουμε στα παλιότερα μοντέλα, αλλά το λόγο έχει η συνάδελφος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, απλώς είναι κρίμα που δεν είναι πολύ παρόντες στην αίθουσα αυτή τη στιγμή, με στη μέρα. Κρίμα που δεν ακούν ε, αυτές τις δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικέ αυτέ οι παρουσιάσει για τις μετέπειτα συζητήσεις μας. Τελικά βλέπουμε ότι η Βαλτική θάλασσα δεν γίνεται αντιληπτή ω μια από τι θάλασσες με τη μεγαλύτερη ρήπανση, παρόλο που ισχύει αυτό. Ακούσαμε ότι γίνεται με τα απόβλητα, με την ε, ρήπανση από τη Γεωργία δευτερογενή ρήπανση ή φαινόμενα ρήπανσης. Αργούν να εκδηλωθούν αλλά εκδηλώνονται. Όλα τα πολίματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τον Nord Stream, ο αγωγός αυτός αναφέρθηκε. Μιλήσατε για τον πόνους Όλα αυτά μας ανησυχούν. Τα αριθμητικά στοιχεία ιδίως μας ανησυχούν πολύ. Οι επιστήμονες έχουν ε, διαπιστώσει ότι η οξικότητα, η οξύτητα μάλλον συνολικά έχει αυξηθεί πολύ ιδίως στα χαμηλότερα στρώματα, και γιατί ο πυθμένας της θάλασσας έχει επιδείνωση στις ε, συνθήκες του λόγω των εκρηκτικών που ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται στην Αλία ή κάποιες φορές να μην ακολουθήθηκαν οι κανόνες για τις περιπτώσεις αγωγών όπως το Nord Stream λόγου χάρη. Ίσως όλοι αυτοί οι παράγοντες να είναι αλληλένδετοι. Και το αποτέλεσμα είναι προγράμματα όπως το Bonus ε, ή το Balto για την Αλία να απαιτούν μεγαλύτερη συνεργασία ε, και με τις χώρες ε, που βρίσκονται γύρω από την Βαλτική αλλά και με τρίτες χώρες για τις οποίες επίσης ε, δημιουργούνται προβλήματα όπως η Ρωσία ή η Λευκορωσία. Είναι πολλοί επιστήμονες που πραγματικά ανησυχούν διότι η Ρωσία δεν επιτρέπει στους εμπειρογνώμονές μας να κάνουν επιστημονικές δοκιμές στα εθνικά της ύδατα. Στα χώρια ύδατα όμως αυτό δημιουργεί δυσκολίες, ιδίως γιατί υπάρχουν και πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου ανοιχτά του Καλίνιγκρατ. Αυτά λοιπόν ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να περιοριστούν οι ζημιές ε, στη Βαλτική, να προβλεφθεί ένα πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων για τις προκληθήσεις ζημιές. Μας ανησυχεί πολύ το γεγονός ότι στο Καλίνιγκραντ υπάρχει πρόγραμμα για νέο πυρηνικό σταθμό λόγω χάρη θα χρησιμοποιηθούν ε, για το πρόγραμμα αυτό και τα νερά του ποταμού Μάλμα, που είναι ποταμό ο οποίο εκβάλλει στην Βαλτική. Είναι πολλέ οι πηγέ τη ρήπανση, λοιπόν. Εσεί τι γνώμη έχετε, Υπάρχει ε, διασύνθεση των φαινομένων αυτών. Η εξόριξη πετρελαίου λόγω χάρη και η κατάσταση του πυθμένα της Βαλτικής. Η κυρία Χάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση έχω για τον κύριο Κνουτήλε και τον κύριο Κούσταυσον κυρίως. Για το πρόγραμμα δράσης Helcom. Στο πρόγραμμα αυτό δράσης του Helcom υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος με λεπτομερή προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία. Αλλά όπως ξέρουμε η Helcom μπορεί να κάνει συστάσεις μόνο, τίποτα άλλο. Τι νομίζετε ότι θα γίνει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέτρα αυτά που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της Helcom γίνουν υποχρεωτικά, δεσμευτικά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει σε νομοθετικές διατάξεις. Ένα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι κλιματικές αλλαγές οδηγούν και σε πιο πολλές βροχοπτώσεις. Και στη Βαλτική θάλασσα λοιπόν. Πριν από 11 χρόνια είχαμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα με πλημμύρες που είχαν γίνει στο ποτάμι Όντρα. με πλημμύρες εξαιτία του Βιντούλα. Η κατάσταση στη Βαλτική θάλασσα λοιπόν μας θυμίζει εκείνη την περίοδο. Αλλά εγώ δεν θέλω να ρωτήσω τόσο για τα ζωτούχα και τα φωσφορικά. Θέλω να ρωτήσω περισσότερο για τα βαρέα μέταλλα και την συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων στη Βαλτική θάλασσα. Ψαρεύουμε πολύ στη Βαλτική θάλασσα και θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν απειλές για την ανθρώπινη υγεία. Ποιος θα απαντήσει πρώτος, ο κύριος Γκούσταυσον. Ναι. Απαντήστε παρακαλώ. Θα απαντήσω εγώ πρώτα γιατί η πρώτη ερώτηση, λέει ο κύριος θα απευθύνθηκε σε μένα. Ίσως να γνωρίζετε, από το 1994-1995 έχει αναθεωρηθεί η κατάσταση όσον ε, αφορά ε, πυρομαχικά που έχουν βρεθεί στη Βαλτική θάλασσα. Σε σχέση με το πρόγραμμα Nord Stream, απλώς και μόνο για να δούμε λιγάκι την τύχη που περιμένει τα τοξικά στα βάθη της Βαλτικής θάλασσας, με το HELCOM έχουμε ξεκινήσει ένα νέο σώμα το οποίο εξετάζει και αναθεωρεί τις πληροφορίες που έχουμε βάσει των ε, τελευταίων μας ε, δεδομένων. Τέλη της χρονιάς θα έχουμε έκθεση από την ομάδα αυτή στη Helcom. Η Πολωνία έχει ηγετικό ρόλο, ρόλο σε αυτή τη δουλειά. Τώρα όσον αφορά τον έλεγχο και τους φόβους και τις ανησυχίες για το ότι η Ρωσία δεν δίνει στοιχεία και δεν επιτρέπει τον έλεγχο ούτε επιτρέπει επιστήμονες από άλλες χώρες να πάνε και να μετρήσουν το βαθμό ρήπανσης της Βαλτικής θάλασσας στα δικά τους χωρικά ύδατα, πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά το Καλίνικραντ έχουμε πολύ καλύτερη συνεργασία τώρα. Έχουμε αρκετές πληροφορίες για να ελέγξουμε την κατάσταση στη Βαλτική θάλασσα και για να κάνουμε αυτήν την ε, ολιστική αξιολόγηση στην οποία αναφέρθηκα πριν. Ξέρω ότι οι Εστονοί και οι Φιλανδοί συνάδελφοι και αυτοί συνεργάζονται με την Αγία Πετρούπολη και με επιστήμονες από εκεί και παίρνουν πολλές πληροφορίες για τον έλεγχο των υδάτων. Τώρα, για νέο πυρηνικό σταθμό στο Καλίνιγραντ και τη θέση της Helcom Μα δεν είναι μόνο το Καλίνικραντ και δεν είναι και μόνο η Ρωσία όπου γίνεται σχεδιασμός και κατάσταση νέων πυρηνικών σταθμών. Υπάρχουν διάφορες χώρες που αναπτύσσουν αυτό το είδος ενέργειας. Αλλά και πάλι υπάρχει διαφορετικό σώμα εργασίας στο HELCOM που ασχολείται με τέτοιες δραστηριότητες. Κοιτάμε λοιπόν από κοντά τι δραστηριότητες υπάρχουν ήδη, τι σχέδια υπάρχουν και ανάλογα κάνουμε προτάσεις. Θέλω να απαντήσω επίσης στο σχόλιο της κυρίας Χάση για τη γεωργία και τα σχετικά μέτρα στην Βαλτική παρόλο που η ερώτηση δεν απευθύνθηκε σε μένα αλλά περισσότερο στους κύριους Κνούτιλα και Γκούσταυσον. Πάντως για το Βαλτικό τμήμα δεν έχουμε μόνο συστάσεις, έχουμε και κάποιες νομικές υποχρεώσεις για μέτρα στη Γεωργία. Υπάρχει το τροποποιημένο παράρτημα 3 της εθήκης του Ελσίνκη που αναφέρεται σε νομική υποχρέωση που έχουν όλα τα συμβαλόμενα μέρη για την πρόληψη της μόλυνσης από την Γεωργία. Υπάρχουν όμως και άλλα μέτρα που εφαρμόζονται στην Γεωργία ανάλογα με τις προϋποθέσεις, με τις συνθήκες, εδάφους κλπ. καθορίζονται αυτές. Τέλος, Πρόεδρε, για τα βαρέα μέταλλα. Ίσως ο Σέπο Κνούτιλα να μπορεί να απαντήσει καλύτερα, αλλά γενικά μιλώντας θα έλεγα ότι ανεξάρτητα από τις πλημμύρες, ανεξάρτητα από τις κλιματικές αλλαγές, η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων, των παραδοσιακών, στη Βαλτική, υδράργυρος, κάδμιο, μόλιβδος κλπ. μειώνονται. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μας για την ασφάλεια των τροφίμων. Σήμερα το πρωί θα ακούσατε για τις διοξίνες στα λιπαρά ψάρια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία θα έλεγα από τα βαρέα μέταλλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κουστάφσον. Όπως είπα, λέει ο κύριος Κνουτίλα, οι απορροές από τη Γεωργία αποδείχθηκαν δύσκολες να μειωθούν. Και στην βάση της εμπειρίας που έχουμε στη Φιλανδία, όπου μειώσαμε τις ποσότητες τεχνητών λιπασμάτων για τον φόσφορο τουλάχιστον στο 1 τρίτο παρόλα αυτά δεν βλέπουμε καθαρή μείωση στην επιβάρυνση από απορροές της γεωργίας. Παρόλο που εφαρμόζουμε πολλά μέτρα για να μειώσουμε την επιβάρυνση από τη γεωργία, Φαίνεται ότι χρειάζεται να περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα πριν να δούμε αποτελέσματα. Μέχρι ότου να δούμε αποτελέσματα μάλλον. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι ε, δεν πρέπει να λάβουμε τα μέτρα αυτά. Αντιθέτως, πρέπει να αρχίσουμε να, να επιβάλλουμε όλα τα δυνατά μέτρα για να μειώσουμε την επιβάρυνση από τη γεωργία της Βαλτικής εάν θέλουμε να μειώσουμε τη συνολική επιβάρυνση εν τέλει όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για τη Βαλτική θάλασσα. Πρέπει να μειώσουμε λοιπόν μέχρι το 2021 κατά 50.000 τόνους το, το, το άζωτο και αυτό μπορεί να γίνει με βελτίωση των ε, μηχανισμών καθαρισμού των υδάτων. Το μισό από αυτό είναι από τη Γεωργία. Έχει λοιπόν τεράστια επιρροή ο γεωργικός τομέας, αλλά ίσως αλλά θα δούμε τέλο πάντων. Για τα βαρέα μέταλλα συμφωνώ με τον συνάδελφό μου κύριο Τούρκιν που είπε ότι αντί για τα βαρέα μέταλλα πιο πολύ εγώ θα ανησυχούσα από άλλα θέματα, από, άλλα, από άλλες ουσίες, για παράδειγμα ορμόνες, για παράδειγμα κατάλοιπα ναρκωτικών ουσιών, από χημικά κοινή χρήση των οικοκυριών που χρησιμοποιούνται καθημερινά και που καταλήγουν και περνούν μέσα από τις εγκαταστάσεις ε, καθαρισμού των οικιακών αποβλήτων που δεν συγκρατούν τα χημικά αυτά. Άρα πρέπει να μειωθεί η χρήση τους. Πρέπει να περιοριστεί η χρήση τους στην πηγή η επεξεργασία των υδάτων δεν αρκεί. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν οικιακών αποβλήτων είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο ενισχυτικός από τα βαριά μέταλλα σήμερα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας, ο κ. Γκούσταυσον. Yes, I, I, I just uh, Απλώς να πω κι εγώ ότι όταν είδα τις αυξήσεις στην ε, παρουσία αλγών στην Βαλτική, κατάλαβα ότι δεν είχαν καμία σχέση με το πρόγραμμά μας, διότι εδώ υπήρχε μια συνολική τάση σε ολόκληρη τη Βαλτική. Δεν ήταν ε, άμεση διασύνδεση. Τώρα, εάν από την οικοδόμηση αυτή που αναφέρατε και τι σχετικές δραστηριότητε, υπάρχει αντίκτυπο στη Βαλτική, δεν ξέρω γιατί δεν παρακολουθούμε συγκεκριμένα εργοτάξια και την, ε, τον αντίκτυπό τους. Νομίζω ότι θα ήταν σωστό να παρακολουθούνται με, με λεπτομέρεια τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες σίγουρα έχουν επιπτώσει στο περιβάλλον. Να προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος τώρα της ακροάσεως. Πώς να μειωθεί δηλαδή ο ευτροφισμός από την γεωργία στη Βαλτική. Εδώ έχουμε δύο πανελίστ, την κυρία Δίθα Πιέτοβα κυρία Πιετοβά είναι της Κεντρικής Ενώσεως Γεωργικών Παραγωγών και Ιδιοκτητών Δασών. Και ο καθηγητής κύριος Γκράνστετ στο Ινστιτούτο Βιοδυναμικής Project. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή σας που με προσκάλεσε να σας κάνω αυτή την ομιλία. Η ομιλία αυτή απηχεί τα σχόλια των γεωργών αλλά και των ε, επιστημόνων. Εδώ μας ενδιαφέρει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τον περιορισμό των απορροών από τη γεωργία. Χρειαζόμαστε βιώσιμε γεωργικέ πρακτικές που να επιτρέπουν την παραγωγή τροφίμων. Υψηλή παραγωγικότητα, καλύπτοντας το περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα και την έκκληση θρεπτικών συστατικών ε, στη θάλασσα. Δύο βασικοί τομείς όπου η γεωργία έχει δυνατότητα να βελτιωθεί περαιτέρω προς τις οικολογικές της αποδόσεις και να βελτιωθεί και η οικολογική κατάσταση της Βαλτικής είναι η εξή. Ο έλεγχος της διάβρωσης από τα καλλιεργούμενα εδάφη, έπειτα η καλύτερη λίπανση των εδαφών με αποτελεσματική χρήση και ορυκτών και οργανικών λιπασμάτων συμπεριλαμβανομένης της κόπρου και τρίτον η διαχείριση της άρδευσης ε, σε σχέση με τα σιδάτινους δρόμους και τα καλλιεργούμενα εδάφη. Εάν δούμε λεπτομερώς τα μέτρα αυτά πρέπει να θυμηθούμε κάποιες βασικές ιδέες για την καλλιέργεια, τη γεωργία. Να θυμόμαστε ότι τα, οικοσύστημα, τα οικοσυστήματα των καλλιεργούμενων γεών δημιουργούν πάντοτε ένα ευρύτερο οικοσύστημα που επηρεάζεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητε. Σε προκειμένου να παράγουμε τρόφιμα πρέπει να αγγίξουμε το έδαφος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος, την επιφάνεια του εδάφους για την υποδοχή των σπόρων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει παρουσία μικροβίων και οργανικών ουσιών. Εδώ υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για διαρροή αζότου αλλά μπορεί και το άζωτο να φτάσει στα φυτά καθώς μεγαλώνει από βιομάζα. Έπειτα, κατά την εποχή της συγκομιδής υπάρχουν ε, πρακτικές όπως η μηχανική συγκομιδή. Αυτά αποδυναμώνουν περαιτέρω το έδαφος δημιουργούνται χημικές ενώσεις που κάνουν πιο ευάλωτο το έδαφος στην διάβρωση. Αυτό σημαίνει απώλεια εδάφους από την χρήση του νερού και τις καιρικέ συνθήκες. Διάβρωση σημαίνει περισσότερο φόσφορο και άζωτο που μεταφέρονται μαζί με τα μόρια εδάφους. Οι απορροές, οι γεωργικές απορροές στη Βαλτική από τις γεωργικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν και με την αποστράγγιξη των υδάτων, των εσωτερικών υδάτων. Αυτό οφείλεται στις χερικές συνθήκες. Η απώλεια συστατικών, θρεπτικών συστατικών προς τη θάλασσα είναι ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Επειδή υπάρχουν φαινόμενα όπως οι ισχυρές βροχοπτώσεις, τα οποία είναι όλο και πιο συχνά. Στις περισσότερες περιπτώσεις η έκκληση των θρεπτικών συστατικών κατά την περιοχή, κατά την περίοδο μάλλον ε, άνθησης των φυτών ε, είναι μικρότερη. Στην άνοιξη το φθινόπωρο ε, είναι περιορισμένη η απορροή από ότι το χειμώνα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Το χειμώνα είχαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα στη Φιλανδία, ακριβώς εξαιτία της διάβρωσης του εδάφους και της μεταφοράς μορίων εδάφους. Πώς να ελέγξουμε όμως τη διάβρωση. Πώς να προστατεύσουμε τα εδάφη μας πώς να ελαχιστοποιήσουμε την αποστράγγιξη και τη μεταφορά των μορίων εδάφους τα καλλιεργούμενα εδάφη και τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να παραμείνουν στην καλλιεργούμενη γη. Παρά τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων ε, που περιέχουν άζωτο, όπως είπε και ο Δ. Κνούτιλα προηγουμένως, δεν έχουμε μπορέσει να αναχαιτήσουμε πλήρως την αποστράγγιξη. Οι απώλειες φωσφόρου είναι περίπου ένα κιλό ανακαλλιεργούμενο εκτάριο έδαφος. εδάφος και αυτό δίνει μεγάλε ποσότητε φωσφόρου. ο επαρκή έλεγχο λοιπόν τη διάβρωση σημαίνει ε, έδαφος το οποίο δεν έχει αποδυναμωθεί και είναι ισχυρό. Επιτρέπει την απορρόφηση των υδάτων εντός του εδάφους χωρίς να αποσπώνται μόρια. Άρα η δομή, η διάρθρωση του, είδους, του, του ίδιου του εδάφους είναι σημαντική. Οργανικές ύλες και μακροβιολογικές, μακροβακτηριολογικές δραστηριότητες μπορούν να λάβουν χώρα σε ένα τέτοιο πλούσιο έδαφος. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για όλες τις ε, γεωργικές δραστηριότητες. Έπειτα, ο Τη διάβρωση. σημαίνει ότι μετά τη συγκομιδή θα πρέπει να προστατεύονται τα εδάφη από τα κατάλοιπα και να υπάρχει αμέσως νέα καλλιέργεια, ώστε το δυνατόν συντομότερα. Υπάρχουν πρέπει να προωθηθούν πρακτικές που επιτρέπουν τον έλεγχο της διάβρωσης και να μένει το έδαφος στη θέση του η φύτευση ε, φυτών και καλλιεργειών στο μήκος των υδάτινων πόρων επιτρέπει την ε, διατήρηση του εδάφου στη θέση του και βελτιώνει τη βιοπικιλότητα καθώς και το τοπίο, ε, το οικολογικό τοπίο. Υπάρχουν και χημικά μέτρα που μπορούν να επηρεάσουν τη δομή του εδάφους. Ο γύψος που αυξάνει την ηλεκτρική αγωγημότητα του εδάφους μπορεί να μειώσει την διάβρωση του εδάφους και την απώλεια σε φόσφορο κατά 60%. Ας περάσουμε όμως τώρα στη χρήση των λιπασμάτων ε, που έχει σχέση με τον έλεγχο της διάβρωσης. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην καλύτερη ετικετοθεσία, τις τεχνολογικές τη χρήση των τεχνολογιών και τις πρακτικές, για τη χρήση και των ανόργανων και των ορυκτών λιπασμάτων. Πρέπει να ε, επιδιώξουμε την εφορία και την αποτελεσματικότητα των λυσμασμάτων τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται στο καλύτερο δυνατό σημείο, κάτω από την επιφάνεια του εδάφου, στην καλύτερη χρονική στιγμή και για τους καλύτερους σκοπούς. Το επίπεδο της ε, προέλευσης των ε, θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ακριβώ για την καλή ανάπτυξη των φυτών. Τα θρεπτικά συστατικά που θα, θα προέρχονται από τα λοιπάσματα δεν πρέπει να διασπούν την ε, δομή του εδάφους. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν κατάλληλες ε, ετικέτες για τις οργανικές πηγές και για τη μακροβιολογική δραστηριότητα των λοιπασμάτων. Αυτό επηρεάζεται και τι καιρικέ συνθήκε. Επί τη αρχή, λοιπόν, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανόργανων και κλασικών μεθόδων καλλιέργεια σε σχέση με την διαρροή θρεπτικών συστατικών από μια συγκεκριμένη επιφάνεια. Η κατάλληλη στιγμή της εναπόθεσης των λοιπασμάτων με τις κατάλληλες ετικέτες είναι ύψης της σημασίας. Όταν υπάρχει καλή διαχείριση των γεωργικών δραστηριοτήτων, η κλασική γεωργία είναι ακόμη λιγότερο επικίνδυνη για την καλή ποιότητα των υδάτων, όπω και βεβαίω τα καλύτερα, πλουσιότερα εδάφη επιτρέπουν την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών. Ιδίω η διαχείριση του φωσφόρου είναι σημαντική για να έχουμε έγκαιρη ανάπτυξη των φυτών με ένα καλύτερο αποτέλεσμα γεωργικό. Τα, η έντονη χρήση φωσφόρου νωρίς θα αποδυναμώσει τα ε, προϊόντα πριν τη στιγμή της συγκομιδής. Πρέπει λοιπόν το δυναμικό ανάπτυξης να το προβλέψουμε τη στιγμή της σποράς. Αυτό ε, έχει να κάνει και με, τον, με το άζωτο ιδιαίτερος, το οποίο χρειάζεται στο τέλος της, ε, του κύκλου ανάπτυξης. Τα φυτά χρησιμοποιούνται βασικά στοιχεία όπως το φόσφορο και το άζωτο. Οι περιορισμοί όμως τα ποσά που απαιτούν τα φυτά μόνο για την ανάπτυξή τους και όχι για άλλους σκοπούς, βελτιώνουν και μειώνουν τα ποσοστά γενικότερα και των υπόλοιπων θρεπτικών συστατικών και των απορροών τους. Αυτό θα μας επιτρέψει και καλύτερη διαχείριση των εδαφών και αντιμετώπιση των καιρικών συνθήκων. Μια μεγάλη πρόκληση είναι επίσης η ζωική κόπρος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο για να υπάρξει και ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών. Καταγράφουμε την ανάγκη των καλλιεργούμενων φυτών, αλλά η κόπρος κάποιες φορές περιέχει πολύ περισσότερο φόσφορο από ότι άζωτο. Επειδή λοιπόν υπάρχει συσσωρευμένη κόπρος, η συγκέντρωση του φωσφόρου έχει μεγαλώσει στα κτηνοτροφικές μονάδες. Και ε, το θείο ή το άζωτο μπορεί να οδηγούν σε περισσότερη έκκληση φωσφόρου. Αυτό λοιπόν δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Πρέπει να γίνεται η λίπανση σε ποσοστά που να καλύπτουν μόνο τι ζωτικέ ανάγκε των φυτών ε, και την απόσπασή του ε, κατά τρόπο κατάλληλο, κατά τη συγκομιδή την ε, ανάγκε της οδειάς. Αυτό λέγεται καλή πρακτική εσοδείας για την καλή διαχείριση των φυτών. Έχουν γίνει πάντως προσπάθειες για να μειωθούν τα κοπάδια ζώνη, ή κτηνοτροφικές μονάδες στο μέγεθός τους. Και πρέπει οι γεωργοί να διατρέχουν μεγαλύτερες εκτάσεις γης για να διασπείρουν την κόπρο κάποιες φορές και με, μηχανικό, με μηχανικά μέσα. Πάντως χρειάζονται αηφόροι γεωργικές πρακτικές. Η ανάγκη αυτή πρέπει να τονιστεί για να έχουμε καλύτερα οικολογικά αποτελέσματα και καλύτερη οικολογική κατάσταση τη Βαλτική. Ας μην ε, αφήσουμε τώρα το τελευταίο κεφάλαιο της παρουσίασης, ε, την διαχείριση των εδαφών στο μήκος των υδάτινων πόρων. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει και με την καλλιέργεια εδαφών ε, κοντά σε υδάτινους πόρους. Πολλές φορές εκεί περιέχεται φόσφορος, άζωτο και αν όμω κανεί ε, πάρει τη βιομάζα πριν το χειμώνα, μπορεί να επηρεάσει την περιεκτικότητα σε άζωτο και φόσφορο, καθώ και την απορροή των συστατικών αυτών προ τη θάλασσα. Χρειάζονται λοιπόν προσπάθειε εξόριση και υπάρχει κόστο για του γεωργού. Όμω, ένα μέτρο θα ήταν λόγου χάρη τα συστήματα ε, οι υπηρεσίε οικοσυστήματο, προστασία του οικοσυστήματο θα μπορούσαν να προσφέρουν οι γεωργοί προ την κοινωνία, εξυπηρετώντα αυτέ τι ανάγκε. Σήμερα οι γεωργοί μπορούν να γίνουν παράγοντα ελέγχου τη διάβρωση των εδαφών, μπορούν να καλύψουν τι ανάγκε συγκομιδή και να ε, μα επιτρέψουν καλύτερε ε, πρακτικέ διαχείριση των εδαφών στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βαλτική θάλασσα. Οι γεωργοί των χωρών της Βαλτικής έχουν αναλάβει ενεργό δράση που έχει οδηγήσει σε δύο προγράμματα για την Βαλτική Γεωργία και την Βαλτική Κόπρο. Εδώ υπάρχει και ένα εγχειρίδιο με βέλτιστε πρακτικέ, χωρί να πλήττεται όμω ανταγωνιστικότητα η παραγωγή τροφίμων. Η Γεωργία, ο Γεωργό και ο σύμβουλό του όλοι βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντό μα. Βρισκόμαστε στην κατεύθυνση βελτίωση τη οικολογική κατάσταση τη Βαλτική, εάν προωθήσουμε την αηφόρο γεωργία. Οι βελτιώσει δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν και όπω υπόθηκε και σήμερα, έχει πολύ μακριά και αργή μνήμη η Βαλτική θάλασσα. Όμω, εάν μειώσουμε τι απορροέ ε, εσωτερικώ ε, για το φόσφορο και το άζωτο ε, και που προκαλούνται από τη γεωργία θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και αν δούμε τι γίνεται με την περιεκτικότητα φωσφόρου στα εδάφια αλλά και την ύπαρξη φωσφόρου, την παρουσία φωσφόρου στα, ε, τις άλγες, τα φύκη ε, της Βαλτικής θάλασσας, θα καταλάβουμε πόσο διαφορετική χρήση μπορεί να έχει η διαθυμική ουστία. Πρέπει να βελτιώσουμε τις γεωργικές μας δραστηριότητε. Η Βαλτική θάλασσα ω περιφέρεια έχει δραματίσει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση του γεωργικού τομέα μας πρέπει πλέον να επικεντρώνονται οι γεωργοί στην καλύτερη και αηφόρο διαχείριση της γεωργίας και για την ε, αποτελεσματικότητα των καλλιεργειών και για την καλή χρήση της βιομάζας. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει σεβασμός για την προσεκτική και συνετή χρήση των θρεπτικών συστατικών με τρόπο όσο γίνεται πιο αισιόδοξο. Πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για τον έλεγχο της διάβρωσης και την αποστράγγιξη από τις καλλιεργούμενες περιοχών. Πρέπει η γεωργία να είναι υπομονετική, καθώς το έδαφος και η γη αντιδρούν πολύ αργά. Επιπλέον, για την πολιτική της Βαλτικής ελπίζω ότι θα έρθουμε σε αυτές τις προτεραιότητες για να δούμε σφαιρικότερα την κατάσταση της Βαλτικής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή βέβαια να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά που περιγράψατε. Τέλος, ο καθηγητής Γκρανστέτ τώρα έχει το λόγο, ο οποίος είναι από το Ινστιτούτο Βιοδυναμικών Ερευνών, το Πέρας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σουηδικά, εφόσον μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές που με προσκάλεσαν εδώ σήμερα. Εδώ στην διαφάνεια βλέπουμε Εδώ λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε το πρόγραμμα Μπέρας. Εγώ είμαι συντονιστής για το πρόγραμμα αυτό το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρηματοδοτείται ουσιαστικά. Η πρώτη φάση ήταν 2003 με 2006 και τώρα είμαστε στο δεύτερο στάδιο 2010-2013. Η δουλειά μας βασίζεται στην αρχή που λέει ότι η γεωργία είναι η φυσική μας πόρη για το μέλλον. Πρέπει δηλαδή ο κόσμος να μπορεί να ζει από τη γεωργία χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και οι ροές ε, συστατικών να είναι ελεγχόμενες έτσι ώστε να σεβόμαστε τις πηγές και την βιοπικιλότητα. Ε, το πράσινο κομμάτι είναι αυτό που καταναλώνει η γεωργία με την ηλιακή ενέργεια, ενώ το κόκκινο είναι η χρήση της ενέργειας. Η χρήση που κάνουμε εμείς. Σήμερα λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η χρήση είναι πιο σημαντική από την παραγωγή, δηλαδή καταναλώνουμε περισσότερο από αυτά που μπορούμε να παράγουμε με δύο Η Γεωργία σήμερα χρησιμοποιεί περισσότερα ε, ορυκτά από όσα παράγει. Στερεά καύσιμα δηλαδή. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει. Η εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων όπως είναι η βιομάζα μπορεί να βοηθήσει. Η γη θα πρέπει να είναι σε θέση να θρέψει περισσότερο κόσμο και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε την ηλιακή ενέργεια. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό χρειάζονται όμως νέες γεωργικές πρακτικές. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου χρησιμοποιούμε πάρα πολλά στερεά καύσιμα για να σταθεροποιήσουμε το άζωτο και για να χρησιμοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια στη φωτοσύνθεση. Στην Σουηδία έχουμε μια αύξηση από το 50 μέχρι το 85 περνάμε από 21 σε 80 κιλά το εκτάριο. Η διαφορά που βλέπετε ανάμεσα στην κόκκινη και την πράσινη γραμμή είναι πολύ μεγάλη και οφείλεται στο άζωτο το οποίο βρίσκουμε στα τρόφιμα. Αυτό είναι που λέμε ε, το φορτίο που φέρει η Βαλτική θάλασσα. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε τη συνολική εικόνα. Βλέπουμε ότι έχουμε μια σταθεροποίηση όσον αφορά το άζωτο ανάμεσα στο 1980 και 1990 Και έχουμε από την άλλη μία μείωση μετά το 1995. Έχουμε την παραγωγή πρωτεϊνών, ζωοτροφών. Έχουμε αύξηση τελικά των χημικών προϊόντων. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, Οι υπολογισμοί που έχουν γίνει μας οδηγούν στα συμπεράσματα αυτά. Η μείωση τώρα από την άλλη μεριά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό έχει να κάνει με την αύξηση της βιολογικής γεωργίας. 20% επιπλέον επιφάνεια καλλιεργείται βιολογικά στη Σουηδία. Όμως, η αύξηση που είχαμε από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 80 προέρχεται, και το είπε ο κύριος Κνουτήλα ξεκάθαρα, από το ότι διαχωρίσαμε τις γεωργικές καλλιέργειες που επικεντρώνονται στις ζωοτροφές με πολύ φόσφορο κλπ. Και την κτηνοτροφία από την άλλη. Έτσι, παράγουμε ζωοτροφές που απαιτούν μεγάλη επιφάνεια. διαπιστώνουμε ότι ο κύκλος αυτός θεωρήθηκε αποτελεσματικός για τη Γεωργία. Βλέπουμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε ότι το άζωτο που παράγεται στη συνέχεια χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφία, πηγαίνει στην κτηνοτροφία. Εκεί ενσωματώνεται. Υπάρχουν στατιστικά δεδομένα, έχουμε κάνει μελέτες σε 200 ε, εκτροφικές μονάδες και καταλήξαμε σε 230 κιλά εκτάριο τα οποία ε, κίνονται. Δηλαδή επιπλέον άζωτο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. διαπιστώνουμε ότι έτσι δημιουργείται περισσότερο άζωτο εξαιτία της εντατική κτηνοτροφίας, κάτι το οποίο οδηγεί και σε διάβρωση του εδάφους. Φιλανδοί ερευνητέ απέδειξαν ότι ισχύει αυτό, αυτός ο κύκλος. Και εδώ δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στην κτηνοτροφία, Υπάρχει ένα φαινόμενο συγκέντρωσης σε ορισμένες περιοχές στη Σουηδία και τη Φιλανδία και όχι μόνο, και στις άλλες χώρες της Βαλτικής. Εξαρτιόμαστε κατά πολύ από την παραγωγή σιτηρών και από την εξαγωγή τους. Ουσιαστικά δεν πρέπει να έχουμε παραπάνω κεφαλές ζώων από αυτά τα οποία μπορούμε να θρέψουμε ανάλογα με τον χώρο που έχουμε στη διάθεσή μας. Στις χώρες της Βαλτικής, γύρω από τη Βαλτική θάλασσα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πλεόνασμα αζότου, κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε μεγάλες δυσκολίες προκειμένου να διοχετευτεί τελικά το άζωτο στην διαθέσιμη επιφάνεια που έχουμε. Από τις μελέτες μας καταφέραμε να παρακολουθήσουμε την ισορροπία θρεπτικών συστατικών και να μελετήσουμε και την ενεργειακή ισορροπία. Προσπαθούμε ακριβώς να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και την ε, έκκληση. Πρέπει να δούμε ένα παράδειγμα μέτρων. Πρέπει να συγκρίνουμε επίσης την κατάσταση όσον αφορά την ε, βιολογική γεωργία, να δούμε τι διαφορές υπάρχουν. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε 70% λιγότερο πλεόνασμα στην μη συμβατική γεωργία. Έχουμε μία εντατική γεωργία και στην Σουηδία και στη Φιλανδία και μία εντατική γεωργία στην Πολωνία. Εάν η πολωνική γεωργία ήταν εντατική όσο και στη Σουηδία, αυτό θα δημιουργούσε τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ροή των νοσιών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου. Πρέπει να δούμε το σύνολο δηλαδή του κύκλου που λαμβάνει υπόψη την παραγωγή ζωοτροφών και την κτηνοτροφία. Και αυτό μάλιστα βάσει των διαθέσιμων εδαφών. Είναι ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Ecological Recycling Agriculture, ERA. Πρόκειται για μια γεωργία η οποία ανακυκλώνει το σύνολο των συστατικών. Η βιοπικιλότητα γίνεται σεβαστή, προστατεύεται, υπάρχει ισορροπία όσον αφορά τα κοπάδια ανάλογα με την επιφάνεια δηλαδή, και τρέφονται από ζωοτροφές κατά ένα μεγάλο ποσοστό που παράγονται στην ίδια επιφάνεια. Το πρόγραμμα Μπέρας λοιπόν περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους προγράμματα τα οποία μας επιτρέπουν να εφαρμόζουμε τις αρχές αυτές έτσι ώστε να μειώνεται μειώνονται οι ποσότητες οι οποίες ε, καταλήγουν στη Βαλτική θάλασσα. Έχουμε διάφορους εταίρους. Διάφοροι φορείς, καλλιέργειες, τοπικές ε, οργανώσεις συμμετέχουν στα υποπρογράμματα αυτά. Ποιος είναι ο στόχος μας τελικά. Θέλουμε να παράγουμε καλύτερα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή την αρχή της ανακύκλωσης ή εν πάση περιπτώσει του φυσικού κύκλου των συστατικών για να μειώσουμε το φορτίο από τις χημικές ουσίες. Κάποιος πριν το είπε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την βιοπικιλότητα στην Ήπεθρο με τη δράση. Πρώτα απ' όλα έχουμε τους καταναλωτές. Είναι οι καταναλωτές αυτοί που στην ουσία μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν και συζητάμε με πολλούς δήμους και φροντίζουμε ώστε να προμηθεύουμε στα σχολεία, στις καντίνες δηλαδή των σχολείων, οικολογικά προϊόντα. Στη Φιλανδία είδα ε, τις προάλλες ότι οι εταίροι μας στα εστιατόρια του Ελσίνκη ε, χρησιμοποιούν ε, την αρχή της διατροφής για μια καθαρή βαλτική. Και από την άλλη μεριά συμβουλεύουμε τις αρχές σε διάφορα επίπεδα. Έχουμε και ένα πολιτικό μέσο στη διάθεσή μας. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια διαδικασία. Εδώ βλέπετε την τελευταία διαφάνεια. Μπορούμε λοιπόν να λάβουμε δράση στον πολιτικό τομέα. Για να δούμε τελικά τι μηχανισμούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε όθηση σε αυτή την πολιτική διαδικασία που είναι η λήψη πολιτικών αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε ενισχύσει υπέρ της βιολογικής γεωργίας. Υπέρ μιας κτηνοτροφίας προσαρμοσμένης στις ε, ανάγκες. Επίσης φροντίζουμε για επενδύσεις από πλευράς των γεωργών, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποίησαν κακές πρακτικές στο παρελθόν και τώρα περνάνε σε καλύτερες. Έχουμε και την ε, οδηγία που έχει να κάνει με τα υδατά. Θέλουμε στη δράση μας να συμπεριλάβουμε και τις ροές αυτές που καταλήγουν στην Βαλτική από τα ποτάμια. Θέλουμε να μειώσουμε, όπως είπαμε, το φόρτο αζότου που χύνεται στη Βαλτική. Άρα λοιπόν θέλουμε να προωθήσουμε τη γεωργία που βασίζεται στην ανακύκλωση για να μειωθεί η ποσότητα αυτή αζότου. Και πρέπει να τηρείται η αρχή που λέει ότι ο ρηπαίνων πληρώνει. Αυτό είναι και το βασικό θέμα. Θα στοιχήσει βέβαια κάτι παραπάνω σε αυτόν που ρηπαίνει, αλλά πρέπει να γίνει και να πληρώνουν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες ρηπαίνουν και να θαρρύνουμε συγχρόνως έτσι τους γεωργούς να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να μην ρηπαίνουν. Υπάρχει βέβαια και ο νομοθετικός δρόμος. Βάσει της ε, νομοθεσίας σιγά σιγά πρέπει να προσαρμόζεται η κτηνοτροφία. Έπειτα οι πληρωμές πρέπει να γίνονται ανάλογα με τις συνθήκες που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, αν προστατεύουν το περιβάλλον. Με ό,τι πόρους έχουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά για την ενδιαφέρουσα ανάπτυξη του θέματος και ελπίζω οι ιδέες αυτές να βρουν πολλούς υποστηρικτές. Παρ' όλα αυτά, προμηνών όταν εξετάσαμε τον τρόπο μάλλον την μαζική χειροτροφία είχαμε διαπιστώσει πολύ αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής αυτής και έχουμε ορισμένες αμφιβολίες. Ε, φτάνουμε πλέον στο τέλος της ε, ε, ακροάσεως και παρακαλώ κυρία Χάση να συναγάγει τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά όλους τους ομιλητές για το εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο καθώς επίσης ευχαριστώ τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος που διοργάνωσε την ακροασία. ελπίζω να λάβουμε, να λάβει η γραμματεία δηλαδή τις διάφορες ε, παρεμβάσεις ώστε να μπορούμε να τις έχουμε στη διάθεσή μας. Είδαμε νομίζω ε, πιστικές ενδείξεις για τις μεγάλες αλλαγές στη Βαλτική θάλασσα τα τελευταία 100 χρόνια και αλλαγές τις οποίες προκάλεσαν κυρίως οι ανθρώπινες παρεμβάσεις και οι αλλαγές αυτές σε πόλεις, στην Γεωργία κλπ. Νομίζουμε ότι ο στόχος, η στόχη των ανθρώπων ήταν η βελτίωση τη της ζωής των κατοίκων της ε, περιοχής γύρω από την Βαλτική. Η δε μόλυνση της Βαλτικής ήταν μια ε, συνέπεια που δεν ήταν βεβαίως ε, επιδιωκόμενη. Αλλά οφείλουμε να λάβουμε υπόψη σοβαρά το γεγονός ότι η Βαλτική θάλασσα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, ότι είναι από τις πιο ε, μολυσμένες θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο. Θα πρέπει επίσης να δράσουμε σεβόμενοι τις ευθύνες που έχουμε και ε, όπως είπατε και στην αρχή η Βαλτική είναι σχεδόν εσωτερική θάλασσα της Ευρώπης. Άρα η οικολογική της κατάσταση, η περιβαλλοντική της κατάσταση είναι κατά το πλήστον στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ε, που είδαμε ποια, ποιες ήταν οι συνέπειες του διαχωρισμού της ε, κτηνοτροφίας από την παραγωγή σιτηρών. Ποιες ήταν οι συνέπειες δηλαδή για την γεωργική παραγωγή, ποιες ήταν οι συνέπειες για, την, για τις απόρριες ε, τροφικών υλών από τη γεωργία και την κατάληξή τους στην θάλασσα. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα παράδειγμα που δείχνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο, ενώ απαιτούνται σημαντικές αλλαγές. Άρα χρειαζόμαστε, νομίζω, αλλαγή νοοτροπίας, ώστε και τα αστικά κέντρα και η βιομηχανία, αλλά και η γεωργία να γίνουν πιο βιώσιμες, αλλά και ευφιέστερες στην περιοχή γύρω από τη Βαλτική, βέβαια και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Helcom έχει θεσπίσει το σχέδιο δράσης με πολλά επιμέρους σημεία. Ένα από αυτά είναι να Πάψει να χρησιμοποιείται φόσφορο στα απορριπαντικά. Την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή Περιβάλλοντος ψήφισε τη σχετική έκθεση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει σε αυτή την ε, θέσπιση της σύστασης αυτής ως νομικής υποχρώσεως. Υπάρχουν και τα άλλα σημεία του σχεδίου δράσεως της Helcom για την Γεωργία. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να γνωρίζω ή να αποφασίσω ποιες δράσεις θα πρέπει να είναι σε εθελοντική και ποιες σε υποχρεωτική βάση. Πάντως θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την λήψη του σχεδίου δράσεως της Helcom ως ένα είδος εγχειριδίου για το τι απαιτείται να γίνει και στη Γεωργία. Διότι είδαμε ότι και αν ακόμη εκμεταλλευτούμε κάθε δυναμικό που έχουν τα αστικά κέντρα για να μειώσουμε την ευστροφία ή τον ευστροφισμό που ελπίζω να γίνει, πάλι αυτό δεν αρκεί για να θεραπευθεί η Βαλτική θάλασσα. Δεν είναι δυνατόν να βελτιωθεί η κατάσταση στην ε, Βαλτική θάλασσα χωρίς αλλαγές στην γεωργία. Ακούσαμε επίσης ότι η αναθέρμανση του κλίματος καθιστά τις προκλήσεις ακόμα ε, δυσκολότερες και χρειάζεται βέβαια να ξανασκεφτούμε σε βάθος ολόκληρη την γεωργία, ολόκληρη την αγροτική παραγωγή. Το τελευταίο μου θέμα που είναι σχετικό με τις χημικές ουσίες μην λησμονούμε ότι δεν είναι μόνο ο ευτροφισμός, είναι και οι επικίνδυνες χημικές ουσίες που αποτελούν πρόβλημα στη Βαλτική. Για παράδειγμα, όταν συζητεί το η οδηγία REACH για τα χημικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάθαμε ότι κάποια, κάποιες ποσότητες ε, χημικών με σωρευτικό χαρακτήρα που συσσωρεύονται δηλαδή στα ψάρια αλλά και στα πτηνά και στις φώκες ε, της Βαλτικής είναι για παράδειγμα πέντε φορές περισσότερα από ό,τι στην Βόρεια θάλασσα. Χρειαζόμαστε λοιπόν και εδώ δράση. Επίσης πάλι όταν συζητείται εδώ η REACH ένα από τα σημαντικά θέματα που θυμούμε από όλε εκείνε τι συζητήσει, αλλά βέβαια και από το υλικό λόμπι που είχαμε λάβει ήταν ένα μήνυμα που είχαμε λάβει από ε, τοπικές κοινότητες και κυρίως από, τους, ε, από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού των υδάτων και που έλεγαν ότι πολλές από τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στα απόβλητα δεν συγκρατούνται στις εγκαταστάσεις δεν καθαρίζονται δηλαδή τα νερά από τέτοιου είδου χημικές ουσίες. Άρα πρέπει να αφαιρεθούν τα χημικά αυτά, οι χημικές αυτέ ουσίες, πριν να καταλήξουν στου αγωγούς των εγκαταστάσεων καθαρισμού. Και αυτό θα αυξήσει τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε και τους πόρους που έχουμε και για την χρήση των εγκαταστάσεων καθαρισμού των υδάτων, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή ευρύτερα. Άρα τα νερά που θα προκύπτουν μετά τον καθαρισμό θα είναι ευκολότερο να ανακυκλωθούν εάν δεν, εάν δεν περιέχουν πλέον βαρέα μέταλλα αλλά και άλλες ε, επικίνδυνες χημικές ουσίες. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά. Ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους όσοι συμμετέσχουν στην ακρόαση και ελπίζω η ακρόαση να ε, συμβάλλει στο έργο όλων μας για να γίνει η Βαλτική ε, καθαρότερη και υγιέστερη. Ευχαριστούμε κυρία Χάση. Να κηρύξω τη λήξη της συνεδρίασής μας. Επόμενη συνεδρίαση 13 και 14 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ όλους και τους επιρρογνώμονες και τους βουλευτές και τους διερμηνείς και τη συνάδελφο Μορκουνάιτε που έμεινε στο τέλος της ακρόασης.